Ladies and gentlemen, please Καλημέρα κυρίες και κύριοι, λέει η Πρόεδρος. Αρχίζει η συνεδρίαση της Υποεπιτροπής για Ασφάλεια και Άμυνα. Πρέπει να σας ενημερώσω για τη συνεδρίασή μας το εξή, ότι μεταδίδεται από το ίντερνετ, στο ίντερνετ, και έχουμε εξασφαλίσει ε, διερμηνία για τέσσερις ε, συναδέλφους της Επιτροπής μας. Τώρα, να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αντίρρηση, οπότε εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιος να ζητεί το λόγο σχετικά. Οπότε πάμε στο επόμενο σημείο της διατάξεως που είναι η ανταλλαγή απόψεων. Με τους ε, εξέχοντες καλεσμένους μας. Έχουμε τρεις προσκεκλημένους. Το, το, το θέμα μας είναι ο υβριδικός πόλεμος, απειλές και προκλήσεις. Και με μεγάλη μου χαρά καλώς όρισε ο Τίμο Κώστερ, ο οποίος είναι διευθυντής στο ΝΑΤΟ για θέματα πολιτικής άμυνας και ε, δυνατοτήτων άμυνας. Επίσης ο κύριος Γκάμπορ Ήκλοντι από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Είναι παλιός μας γνωστός και ο Άιρες Ρικβέλης που είναι σύμβουλος σε θέματα αμήνης και υπηρετεί στην ε, λετονική αντιπροσωπεία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Θερμά καλωσορίσματα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα ο υβριδικός πόλεμος. Είναι κάτι το οποίο που ήρθε στην επικαιρότητα μετά την ε, ρωσική εισβολή στην ε, ε, Ουκρανία μετά την παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας. Αλλά παρόμοια φαινόμενα έχουμε παρατηρήσει και αλλού. Βλέπουμε ότι όλα αυτά είναι προκλήσεις και αφορούν την ασφάλειά μας και αυτές οι άλλες προκλήσεις αφορούν το Ισλαμικό κράτος. Οπότε χωρίς να πούμε τίποτε άλλο να δώσουμε τη σκητάλη στον πρώτο από τους καλεσμένους μας. Τον Τίμο Κώστερ. Κύριε Διευθυντά, έχετε το λόγο. Τίμο. Thank you. Um, <clears throat> good morning, ladies Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. thank, uh, Miss... Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την Πρόεδρο κυρία Φωτίνγκα και θέλω να εκφράσω και τη χαρά μου για τη συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση. Το θέμα του υβριδικού πολέμου είναι κάτι που ενδιαφέρει και την Ένωση και το ΝΑΤΟ. Το Εθνικό Κοινοβούλιο και τα εθνικά τι αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο για την ενίσχυση των προσπαθειών για καλύτερη άμυνα και ασφάλεια και αυτό έχει πολλές απόψεις και υβριδικές απειλές και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φυσικά θέλει να συμβάλλει στην ε, βελτίωση αυτών των μεθόδων άμυνας. Οι επιθετικές δραστηριότητες της Ρωσίας στην Ουκρανία τόνισαν ποιες είναι οι απειλές που αντιμετωπίζουμε και με αυτή την ευκαιρία δημιουργήθηκε η έννοια της υβριδικής στρατηγικής. και το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος χρησιμοποιεί υβριδικό πόλεμο, δηλαδή στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα. Το ΝΑΤΟ και η Ένωση μπορούν, μόνο από μπορούν καλύτερα από κοινού να αντιμετωπίσουν τέτοια απειλή. Πρέπει να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιούμε όλα μας τα μέσα και διπλωματικά και χρηματοδοτικά και πληροφοριακά και στρατιωτικά και όλα. στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ουαλία τονίστηκε η ανάγκη η συμμαχία να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τέτοιου είδους απειλές. Και το Φεβρουάριο, τον περισμένο Φεβρουάριο, η Υπουργεία Αμήνης των χωρών του ΝΑΤΟ θέλησε να δημιουργηθεί μια στρατηγική, νατοϊκή στρατηγική αντιμετώπισης υβριδικών πολέμων και απειλών. όπως θα πει και ο Γάβος Ινκλόντι, η Ένωση επίσης επεξεργάζεται την ανταπόκρισή της στις υβριδικές απειλές. Α, εδώ πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία νομίζω. Η... Το ΝΑΤΟ έχει το προτέρημα να αναλαμβάνει τη στρατιωτικό σκέλος των... της αντιμετώπισης και η Ένωση την πολιτική, οικονομική και μη στρατιωτική μέθοδο ή και εργαλεία. Θα έλεγα λοιπόν ότι έχουμε συμπληρωματικούς ρόλους και πρέπει να διασφαλίσουμε συνεπή συνδυασμό των προσπαθειών μας. Η στρατηγική λοιπόν που επεξεργάζεται το ΝΑΤΟ, για να σας πω τι λέει, θέλει να περιγράψει πρώτον τι είναι το υβριδικός πόλεμος και δεύτερον πώς αντιμετωπίζεται και ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του ΝΑΤΟ. Υπάρχει λοιπόν ρόλος και για άλλους, για μεμονωμένα κράτη και για άλλους διεθνείς οργανισμούς. Ζωτικό στοιχείο της στρατηγικής μας θα είναι η διατύπωση του τρόπου με τον οποίο το ΝΑΤΟ θα συνδυάσει τις δραστηριότητες τους με δραστηριότητες του με δραστηριότητες άλλων. Βέβαια το έθνος που γίνεται θύμα επίθεσης είναι ο κύριος υπεύθυνο για την αντιμετώπιση. Ας πούμε η υπονόμευση είναι θέμα εσωτερικής ασφαλείας του κράτους. Αλλά από την άποψη του ΝΑΤΟ μπορεί το σύμμαχο κράτος να ζητήσει την ανάπτυξη ειδικών δυνάμεων από τη συμμαχία. Μπορεί να στραφεί και προς την Ένωση για να ζητήσει βοήθεια για συνοριακούς ελέγχους ή αστυνόμευση. Γενικά η στρατηγική θέλει να απομυθοποιήσει το υβριδι, τον υβριδικό πόλεμο. Δεν είναι κάτι τελείως καινούριο. Είναι μια προέκταση των κλασικών μεθόδων επίθεσης και πολέμου. Αλλά στο σημερινό κόσμο υπάρχουν απλώς και νέες εξελίξεις που προσθέτουν νέες, νέα στοιχεία κινδύνου. Ας πούμε, μερικά από αυτά είναι τεχνολογικά κυβερνοεπιθέσεις, ας πούμε. Και μερικά κράτη είναι πιο ευάλωτα σε οικονομική υπονόμευση, αν εξαρτάται ας πούμε ένα κράτος από την προμήθεια αερίου από κάποια χώρα της Ανατολικής Ευρώπης. Um, Και κυρίως οι επικοινωνίες έχουν τεράστιες δυνατότητες εδώ. Η Ρωσία όπως είπαμε λαμβάνει αποφάσεις μονολυθικά όπως το είδαμε και με την Κρυμαία και την Ουκρανία. Και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να παίρνει αποφάσεις επειδή παίρνονται από έναν άνθρωπο πολύ πιο γρήγορα. Ενώ το ΝΑΤΟ και η Ένωση είναι δημοκρατικοί οργανισμοί και βασίζονται σε κανόνες. Uh, we, do not have democracy slow. Δεν πρέπει φυσικά η δημοκρατία να μας καθυστερεί. Δεν πρέπει. Και η ταχύτητα της λήψης αποφάσεων 28 κρατών, κοινοβουλίων, πρωτευουσών κτλ. είναι κάτι ουσιώδες. Ε, ένα στοιχείο της νατοικής ανταπόκρισης μπορεί να κινητοποιηθεί σε 48 ώρες αλλά αλλά μπορεί να ληφθεί η απόφαση της κινητοποίησης το ίδιο γρήγορα. Δεν μπορεί. Η ταχύτητα λοιπόν είναι θέμα πολύ σοβαρό. Δεν είναι μόνο θέμα μετακίνησης δυνάμεων αλλά και η γρήγορης λήψης αποφάσεων με βάση ορισμένους δείκτες, πληροφορίες και μηχανισμούς αλλά χρειάζεται και πρόορος σχεδιασμός βέβαια έγκαιρος. Εμείς βλέπουμε τρεις δυνατές λειτουργίες αντιμετώπισης που είναι προετοιμασία, αποτροπή και άμυνα. Δεν είναι διαδοχικές αυτές οι φάσεις. Η προετοιμασία σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να μπορεί να ταυτίζει απειλές, να τις αναγνωρίζει πολιτικά και να χορηγεί και να απονέμει μάλλον δικαιοδοσίες και ευθύνε. Αυτό βέβαια σημαίνει κατάλληλη συλλογή πληροφοριών καθώς και ασκήσεις. Οι σύμμαχοι πρέπει να ταυτίζουν μόνοι τους τα δύνατα σημεία τους και να βλέπουν τι πρέπει να συμπληρώσουν ή να κάνουν και αυτό σημαντικός ρόλος της Ένωσης τώρα σε αυτό. Τώρα, αποτροπή. Είναι σημαντικό να υπάρχει κυβερνητική προετοιμασία αποτροπής ε, της προσπάθειας κάποιου εχθρού για υβριδική επίθεση. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να μοχλεύσαμε ε, όλα τα μέσα που διαθέτουμε οικονομικά, διπλωματικά, πολιτικά και οικονομικά. Αυτό σημαίνει βέβαια και την ορατή στρατιωτική παρουσία στις συμμαχικές χώρες. Η ετοιμότητα για την στρατιωτική απάντηση είναι κλειδί. Για τους εχθρούς βέβαια, για τους αντιπάλους Το σημαντικό είναι να χρειάζεται ο αντίπαλος να δαπανίσει πολλά για να αντιμετωπίσει την ετοιμότητά μας. Ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπλα όπως διεθνής απομόνωση. Αν αρχίσει μια υβριδική επιχείρηση, φτάνουμε στην έννοια της αμήνης το κράτος υπό επίθεση θα στραφεί σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους ανήκει για να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει και ο ρόλος του ΝΑΤΟ εδώ θα ήταν η ενεργοποίηση των στρατιωτικών του μέσων. Military, and it's Υπάρχουν βέβαια και μη στρατιωτικές οργανώσεις που θα κινητοποιηθούν για να εφαρμοστούν οικονομικές κυρώσεις και πρέπει όλα τα μέσα να συνδυαστούν από κατάλληλο συντονισμό και επικοινωνίες. Το κύριο μήνυμα που θέλω να σας αφήσω είναι ότι με τους τρεις πυλώνες που ανέφερα, δηλαδή προετοιμασία, αποτροπή και άμυνα, όλα αυτά απαιτούν ταχύτητα Ας πω τώρα δύο λόγια για την εσωτερική και εξωτερική διάσταση της στρατηγικής μας. Εσωτερικά μιλάμε για τη δυνατότητα του αρχηγείου του ΝΑΤΟ να παραμένει πλήρως ενήμερο για όλες τις διεθνείς εξελίξεις και να είναι κατά άλλη ε, ικανό να λαμβάνει γρήγορα αποφάσεις. Ο κύριος ρόλος μιας στρατιωτικής συμμαχίας είναι να διασφαλίζει ότι τέτοια υβριδικά σενάρια δεν θα καταλήγουν σε άμεση και κατά μέτωπον στρατιωτική σύγκρουση. Η εξωτερική διάσταση τώρα είναι η ετοιμότητα των συμμάχων και άλλων φιλικών χωρών. Προς το συμφέρον μας είναι να συνεργαζόμαστε με άλλους εταίρους όπως και να είναι ικανοί οι σύμμαχοι αυτοί να αντιμετωπίσουν υβριδικές επιθέσεις. Ανάλογα με τη φύση κάποιου κάθε σενάριου, διαφορετικοί διεθνείς οργανισμοί θα κινητοποιηθούν. Θα κινητοποιούνται. Το ΝΑΤΟ και η Ένωση φυσικά έχουν τους κύριους ρόλους και πρέπει να συνεργάζονται και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι μας πρέπει να είναι η εφαρμογή πρακτικών που θα διευκολύνουν την αμοιβαία κατανόηση του ρόλου του καθενός για την αντιμετώπιση του υβριδικού πολέμου και γρήγορη λήψη αποφάσεων. Τέλος, σε ποιους συγκεκριμένους τομείς θα μπορούσαν να συνεργαστούν το ΝΑΤΟ και η Ένωση. και ο Γκάμπο και εγώ είμαστε σε συνεχή επαφή και εμείς και το προσωπικό μας και ταυτίσαμε τουλάχιστον τέσσερις τομείς, μπορεί και άλλοι να υπάρχουν. Πρώτον, ενημέρωση για την κατάσταση γενικότερα, γιατί και οι δύο οργανώσεις μας πρέπει να έχουν την ίδια κατανόηση και κατανομή ρόλων και απονομή ευθυνών. Γιατί μόνο τότε θα μπορούσαμε να συντονίσουμε δραστηριότητες και αντιδράσεις μας. Δεύτερον, στρατηγική επικοινωνία. Από ό,τι είδαμε και από την Ουκρανία είναι σημαντικό αυτό, αλλά και για το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί τα κοινωνικά μέσα και το ΝΑΤΟ και η Ένωση πρέπει να ενδυναμώσουν την ανάγκη να ανταποκριθούν και σε αυτού του είδους την προπαγάνδα καταλήλως με συντονισμένο τρόπο. Τρίτον, Πολ Στρατ, πολιτική και στρατιωτική συνεργασία. οργάνωση κέντρων διαχείρισης κρίσεων κλπ. που πρέπει να συνεννοούνται τακτικά για να υπάρξει μέγιστη αποτελεσματικότητα. Και τέταρτον, κυβέρ, δηλαδή αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων με εξέταση τρόπων συνδυασμού των συστημάτων μας και κοινών ασκήσεων για να αυξηθεί η δυνατότητά μας αντίστασης και ανταπόκρισης σε τέτοιου είδους επιθέσεις. Δεν είναι βέβαια εξαντλητικός αυτός ο κατάλογος, ακόμα τον επεξεργαζόμαστε, αλλά έτσι για να συνοψίσω. Και οι δύο πλευρές κατανοούν ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας όσο το δυνατόν συντομότερο και από πλευρά του ΝΑΤΟ ο, στόχο, ο στόχος είναι η διάσκεψη του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία το καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ. Oh. Και τώρα ο Διευθυντής CMPD. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καλημέρα σε όλους. Ε, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ. Πάντα χαρά μου είναι. Να έρχομαι εδώ πέρα στην Επιτροπή και να δράσουμε απόψεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να δίνουμε διαφάνεια για το τι κάνουμε, τι προγραμματίζουμε να κάνουμε. Και να ακούμε ποιε είναι οι φιλοδοξίε σας. Προκειμένου να χαράσουμε σωστά την πορεία μας. Χαίρομαι λοιπόν γιατί τρέχουμε εδώ πέρα. Αφού το άκουσα τον Τίμο που κάλυψε μια μεγάλη, ένα μεγάλο τομέα, τόνισε ότι συνεργαζόμαστε πολύ και έχουμε παρόμοιες προσεγγίσεις. Αλλά θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάποια ζητήματα. Καταρχάς, τι εννοούμε υβριδικό και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πω δύο λόγια τώρα για την προσέγγιση στη συνέχεια, την οποία σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δύο λόγια για την διαδικασία του που βρισκόμαστε για να δώσουμε τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τις υβριδικές απειλές, να βοηθήσουμε τα κρατημέλη να είναι καλύτερα προστατευμένα. Και τέλος, ε, ίσως δύο λόγια ως για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως το επιπρόσθετο, το κρασάκι στην τούρτα, αν θέλετε. Τι εννοούμε λοιπόν με τις ευρετικές απειλές. Φυσικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ναι, μιλάμε για ευρετικό πόλεμο και όπλα. Μιλάμε για ευρετικές ε, απειλές. Προτιμούμε τον όρο αυτό. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει ορισμός επίσημος για το τι είναι οι ευρετικές απειλές και δεν πιστεύω ότι χρειάζεται άλλωστε. Όσο καταλαβαίνουμε του τι εννοούμε και τι εύρος θεμάτων αντιμετωπίζουμε στις προσπάθειές μας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό αρκεί. Ποιοι είναι λοιπόν οι βασικοί συντελεστές. Καταρχάς, υπάρχει μια κεντρική ε, οργάνωση και συντονισμό των τακτικών και των μέτρων κατά των εχθρών. Αυτό, όπως ε, είπε και ο Τίμο, δεν είναι κάτι καινούριο. Κοιτώντας ε, τις υβριδικές απειλές, τι εντοπίζουμε, στοιχεία τα οποία είναι ήδη γνωστά. Τίποτα καινούριο λοιπόν. Το μέγεθος όμως, το εύρος της απειλής προέρχεται από το συντονισμό διαφόρων εργαλείων και μέσων που χρησιμοποιεί ο παράγοντας επίθεσης. Αυτό λοιπόν αναγάγει σε διαφορετικό επίπεδο και διαφορετική ποιότητα την απειλή. Καλύπτεται. Πρόκειται για ανοιχτές και, καλυμμένες ε, δραστηριότητες. Περιλαμβάνονται και του ιδίου των δύο ειδών δραστηριότητες. Πρόκειται για στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα επίσης, όπως είδατε περιλαμβάνονται και σκοπός είναι να αποσταθεροποιηθεί το θύμα της επίθεσης. Υπάρχει λοιπόν ε, πάντα ε, ένας ε, συνδυασμός εξαναγκαστικών και μη μέτρων, όπως είδαμε και στη Σερβία. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι συχνά εργάζεται μέσω αντιπροσώπου. Δεν βλέπουμε λοιπόν ε, απαραίτητα τον παράγοντα που κάνει την επίθεση. Αυτό καθιστά ακόμα πιο δύσκολη. Και αυτό φυσικά κρύβει συχνά κρατικούς και μη κρατικούς φορείς πίσω από την επίθεση. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των υβριδικών απειλών είναι ότι πάντα υπάρχει μια μαζική εκστρατεία επικοινωνίας η οποία συνδέεται με τις επιθέσεις αυτές για να υπάρξει μεγαλύτερη αβεβαιότητα για το ποιοι είναι οι πράσινοι, τα πράσινα ανθρωπάκια, ποιοι είναι. Είναι εξωγήινοι, είναι Ρώσοι. Και ο στόχος είναι φυσικά να αυξηθεί η πολιτική επιρροή και η πολιτική υπεροχή σε κάποιες περιπτώσεις σε περιοχές ή και σε χώρες. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι οι βρεδικές απειλές εξελίσσονται και προσαρμόζονται με τον καιρό. Αν, ανάλογα και με τα αντίμετρα τα οποία εισαγάγονται. Γι' αυτό λοιπόν το να προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα σαφή ορισμό του τι είναι η βρετική απειλή δεν θα ήταν μόνο δύσκολο αλλά και αντιπαραγωγικό αν θέλετε ως εγχείρημα. Πρόκειται για μια έννοια η οποία εξελίσσεται και τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται είναι απροσδιορίστα εξορισμού. Το να προσπαθήσουμε λοιπόν να τα περιορίσουμε σε ένα συγκεκριμένο ορισμό ενέχει τον κίνδυνο οτιδήποτε μείνει εκτός ορισμού να μην περιληφθεί στην υβριδική επίθεση, στον ορισμό της. Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οτι μου ανέφερε βέβαια ότι δεν είναι αυτό που βλέπουμε προς Ανατολάς. Οι απειλέ που μας κρατούν ξύπνιους τη νύχτα. Είναι λιγότερο απειλητικά αυτά σύμφωνα με την ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι απειλές από τον Νότο είναι εξίσου σημαντικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν στο μέλλον θα επικεντρωθεί πιο πολύ και από τον ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά τα θέματα ανταπόκρισης στις προκλήσεις που προέρχονται από τον Νότο. Επίσης, η απειλή αυτή είναι εξίσου σημαντική, υπό την έννοια που ότι έχουμε ομολόγους, αν θέλετε, που δεν αντιδρούν απαραίτητα λογικά. Αν υπάρχει λοιπόν ένα ισχυρό, ένας ισχυρός κρατικός ε, φορέας πίσω από μια υβριδική επίθεση, αναμένονται ασφαλώς κάποιες ε, λογικές, ορθολογικές απαντήσεις. Αν όμως κρύβεται πίσω από την επίθεση μια τρομοκρατική οργάνωση, η... ο λογικός χαρακτήρας φθήνει. Θυμάμαι ότι οι συνάδελφοι από την περιοχή του Περσικού κόλπου ανέφεραν συχνά ότι είναι διαφορετική η νοοτροπία που έχουμε στο κεφάλι μας εμείς. Δεν δεχόμαστε μια αμοιβαία επιβλαβή κατάσταση. Αυτά για τον ορισμό. Τώρα, ως προς την ε, προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα κοινό χαρακτηριστικό εντοπίζουμε σε όλες τις υβριδικές επιθέσεις, ότι πάντα στο στόχαστρο είναι οι ευαισθησίες μας, οι ευαλωτότητες μας. Οι μας. Ποτέ δεν ε, είναι στο στόχαστρο τα δυνατά μας σημεία. Εντοπίζουν και ψάχνουν να εντοπίσουν τα σημεία στα οποία είμαστε ευάλωτοι. Αυτό καλύπτει πολλά ζητήματα. Την ενεργειακή εξάρτηση, για παράδειγμα, που ανέφερε ο Τίμο. Ε, οι αδυναμίες μας ε, τις πολιτικές ενσωμάτωσης οι αδυναμίες μας στην ε, πολιτική για το κυβερνοχώρο. Σε υπουργικό επίπεδο μεταξύ των κρατών μέλων προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε την περίπτωση της Ουκρανίας για να δείξουμε ποιες είναι αυτές οι κρίσιμες ευαλωτότητες και τι πεδίο, τι εύρος καλύπτουν. Και εκεί σίγουρα μπορούμε να βρούμε κρίσιμα σημεία σε θέματα διακυβέρνησης, για παράδειγμα, σε θέματα διαφθοράς. Αυτό αποτελεί ένα ευάλωτο σημείο. Ε, έλλειψη εμπιστοσύνης στις δημόσιες αρχές και στις δημόσιες ε, θεσμούς. Ε, μεγάλη εξάρτηση από την ενεργειακή παροχή. Η ύπαρξη μεγάλων πληθυσμών ρωσόφωνων μέσα στην χώρα που θεωρούσαν ότι δεν ε, τύχαιναν τις κατάλληλες μεταχείρισεις. Όλα αυτά αποτελούν ευάλωτα σημεία και νομίζω ότι καταδεικνύουν με σαφήνεια πόσο ευρύ είναι το φάσμα των ευάλωτων αυτών. Το πρώτο βήμα λοιπόν. Για όλους μας. Είναι με σαφήνεια να εντοπίσουμε, να αναγνωρίσουμε ότι όλοι έχουμε ευαίσθητα ευάλωτα σημεία. Όλοι λοιπόν έχουμε ευαίσθητα σημεία τα οποία συχνά έχουμε την αίσθηση ότι δοκιμάζονται. Για παράδειγμα, παραβίαση ενέργειου χώρου. Πράγματα που διαβάζουμε στις εφημερίδες ε, κάθε μέρα. Θα πρέπει λοιπόν να ελέγξουμε πού είναι αυτά τα τροτά μας σε μια... Όλα τα κράτη-μέλη έχουν τέτοια τροτά σημεία. Αυτό είναι σαφές, ακόμα και αν διαφέρουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεσμική ύπαρξη επίσης έχει τροτά σημεία. Οι αποστολές μας μεταξύ άλλων στο εξωτερικό. Και αυτές είναι τροτές. Και κάτι θα πρέπει να κάνουμε προκειμένου να προστατευτούν καλύτερα. Δεδομένου ότι σε κάποιες περιπτώσεις ε, λειτουργούν σε επιθετικά και επικίνδυνα περιβάλλοντα. Και η διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελεί ένα σημείο. Και θα επανέλθω σε αυτό. Αν αποδεχτούμε ότι ένας από τους κρίσιμους στόχους των υπηρετικών ε, επιθέσεων είναι να δημιουργηθεί ασάφεια και βεβαιότητα για το τι συμβαίνει, αν δεν ε, λαμβάνονται οι αποφάσεις σε ένα περιβάλλον αβέβαιο που δεν μας δίνει 100% διασφάλιση και απόδειξη σε κάθε βήμα, θεωρώ ότι αυτό αποτελεί κρίσιμη ευαλωτότητα. Οι αποφάσεις θα πρέπει φυσικά να λαμβάνονται γρήγορα και με αποφασιστικότητα. Αυτό πρέπει να το αποδεχόμαστε. Και οι εταίροι μα έχουν τροτά σημεία και σε κάποιε περιπτώσει είναι πολύ πιο ευάλωτοι και εκτεθειμένοι από ότι και εμεί οι ίδιοι. Και αυτό αποτελεί μια διαφορά μεταξύ της προσέγγισης ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει ουσιαστικά τους εταίρους στο ίδιο επίπεδο. Διαβάζοντας ε, τα βασικά πορίσματα του Συμβουλίου, μας καλούν να εργαστούμε για να καταστήσουμε αντίμετρα για να πετύχουμε καλύτερη προστασία και σε ό,τι αφορά τα κρατημέλη και σε ό,τι αφορά τις χώρες εταίρους. Πολύ ωραία. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να τονίσω και το εξή. Για να υπάρξει καλύτερη προστασία από τι υβριδικέ επιθέσει είναι και θα παραμείνει η εθνική αρμοδιότητα. Κανεί λοιπόν δεν θα πάρει αυτή την αρμοδιότητα από τα κράτη-μέλη, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε το ΝΑΤΟ. Πρόκειται για θέματα εθνικής επικυριαρχίας, πάρα πολύ ευαίσθητα και αυτό πάντα εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Το ερώτημα είναι, όταν πρόκειται για οργανώσει όπως το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι, μπορούν να αποτελέσουν μια καλή πλατφόρμα προκειμένου να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να πετύχουν καλύτερα επίπεδα προστασία μπορούν να παρέχουν πλατφόρμα μέσα από την οποία μπορούν να ενισχυθούν οι εθνικές προσπάθειες. Και εδώ υπάρχουν, θεωρώ, κάποιοι τομείς όπου αυτό είναι ασφαλώς δυνατόν. Η στρατηγική επικοινωνία πάντα αποτελούσε ένα διαπιστωμένο τομέα ενίσχυσης. Το πρώτο βήμα, λοιπόν, είναι να υπάρξει ευαισθητοποίηση και σωστή αντίληψη του τι συμβαίνει, ποιες είναι οι απειλές, ποιες είναι οι στρατιωτικές δράσεις που ενδεχομένως να αποτελούν τμήμα ενός υβριδικού σενάριου. Και για την κατεύθυνση αυτή, ένα από τα βήματα που ακολουθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από εντολή του Συμβουλίου του Μαΐου και του Ιουνίου είναι να δημιουργηθεί ένα κύτταρο σύνδεξης, fusion cell, προκειμένου να συλλέγονται πληροφορίες και μυστικές ε, πληροφορίες που σε μεγάλο βαθμό ήδη υπάρχουν στα κράτη-μέλη προκειμένου να μπορούν τα κατημέλη να βάλουν, αν θέλετε, τα γυαλιά μέσα από τα οποία θα δουν τις υβρετικές επιθέσεις και να συνενώσουν όλες τις πληροφορίες αυτό το Fusion Cell για να έχουμε μια πιο συνολική εικόνα. Ένα άλλο σκέλος της προσπάθειας αυτής είναι το ΝΑΤΟ και το ανέφερε ο, ο Τίμο. Σε μια ιδανική περίπτωση θα πρέπει να δημιουργηθεί μια συνολική κατάσταση προκειμένου να υπάρχει συνολική εικόνα. Και στους δύο οργανισμούς, οπότε θα είναι ευκολότερο να έχουμε συντονισμό των προσπαθειών και να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη σε σχέση με το τι ε, ανταπόκριση θα πρέπει να έχουν. Οπότε για τις ε, κυβερνοαπάντες, αυτό που χρειάζεται, σύνομα για τις ε, κυβερνοαπειλές, θα πρέπει να υπάρχει αντοχή και ανθεκτικότητα. Δηλαδή Εάν έχουμε τέτοιε απειλέ, τα ευάλωτα σημεία μα, τότε εμεί θα πρέπει να μην έχουμε ευάλωτα σημεία. Δηλαδή να μην υπάρχει ε, έδαφος, χώρος, δυνατότητα επίθεση από τον επιτιθέμενο. Οπότε δεν θα πρέπει να έχουμε τέτοια δύνατα σημεία, δύνατους τομείς. Ενέργεια, α πούμε, εκεί να έχουμε ε, διαφοροποίηση όσον αφορά την προμήθεια ενέργειας. Ε, να μην ε, εξαρτώμεθα μόνο από το φυσικό αέριο, ε, να έχουμε υγροπημένο φυσικό αέριο κλπ. Οπότε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να συμφωνήσει αυτή την οδηγία NIS για αυτό το δίκτυο πληροφοριών που αφορούν την ασφάλεια. Ε, επίσης, να αναφέρουμε το, το παράδειγμα της ε, ένταξης της κοινωνίας μας των διαφόρων ε, κοινοτήτων. Να, σε σχέση με την Ουκρανία τι ισχύει. Αντί να αποξενώνει κανείς κάποιες κοινότητες και έτσι να τις κάνει πιο ευάλωτες όσον αφορά την επιρροή του εχθρού, θα πρέπει κανείς να τις αγκαλιάζει, να τις ελκύει, να τους προκαλεί ενδιαφέρον. Να πως πρέπει να αποκρίνεται κανείς. Επίσης, να προσέξουμε και την πρόληψη. Και αυτό είναι πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, αντί κανείς να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις, να τις προλαβαίνει. Κυβερνητική προσέγγιση, όπως είπε ο προλαλής σας. Κάποια από τα κράτη-μέλη, ιδίως η Φιλανδία, Ήδη έχουμε εμπειρία σε αυτό. Άρα μπορούμε να βασιστούμε σε την εμπειρία και να αντιλήσουμε συμπεράσματα. Το επόμενο. Αποτροπή. Αυτό είναι όρο που χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ και γι' αυτό κάποιοι θα πούνε όχι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει τέτοια πράγματα. Ξέρω, ξέρω. Να, τι γίνεται με τις κυρώσεις. Δεν έχουμε τέτοιο ρόλο. Δεν έχουμε στην εργαλειοθήκη μας και την ε, αποτροπή. Για σκεφτείτε καλύτερα. Τι θα πει η αποτροπή. Όχι μόνο να επιδεικνύει κανείς ισχύ ούτω ώστε να αποτρέπει, αλλά το να ε, εφαρμόζει κανείς την αποτροπή ούτως ώστε το όφελος από την επίθεση να ακυρώνεται μέσω αυτής της αντοχής και ανθεκτικότητας. όσον αφορά την απόκριση, ανταπόκριση, για να ολοκληρώσω αυτό το σημείο, να επανέλθω σε αυτό που λέγαμε για την λήψη αποφάσεων. Και αυτό θα πρέπει να γίνεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, οπότε να έχουμε σε πολιτικό επίπεδο αυτή τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων και όλοι επομένως που λάβουν αποφάσεις να καταλάβουν ότι το περιβάλλον ε, όπου χρησιμοποιείται για να παίρνουν αποφάσεις είναι κάτι το αβέβαιο αλλά αυτό δεν είναι λόγος αυτοί να μην λαμβάνουν αποφάσεις Δύο λόγια τώρα για τη διαδικασία στην οποία βρισκόμαστε η εσωτερική προβληματική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις κυβερνοπηλές ξεκίνησε πέρσι, πέρσι το καλοκαίρι πριν τη συνάντηση του ΝΑΤΟ και είχε κληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενώσει τις δυνάμεις της με το ΝΑΤΟ ούτω ώστε να βρεθεί τρόπος κάλυψης αυτών των απειλών. Και μετά έγινε η υπουργική συνάντηση και προέκυψε αυτή η προσέγγιση που σας περιέγραψα και το πιο σημαντικό για μας είναι το Συμβούλιο Εξωτερικών του Μαΐου που μας έδωσε την εντολή να ασχοληθούμε με τις κυβερνό απειλές ή το φρόντι τις υβριδικές απειλές ούτως ώστε η το φραγμα τις υβριδικες απειλες ουτως ωστε η επιτροπη και η υπηρεσία μας φέτος να έχουν ένα κοινό πλαίσιο, κοινή προσέγγιση. Τι θα κάνουμε για τις απειλές αυτές, πώς θα υπάρχει η απαραίτητη ανθεκτικότητα. Και αυτό το σας το τονίζω ιδιαίτερος, γιατί νομίζω είναι ακόμη πιο σημαντικό ούτω ώστε, είπαμε, μέχρι το Δεκεμβρίο φέτος να έχουμε έναν ε, κατάλογο από προτάσεις οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοθούν. Οπότε αυτό είναι το θέμα, όχι να βρούμε μια καινούργια στρατηγική και όλα αυτά τα οποία είχαμε στο παρελθόν να τα βάλουμε στο χρονοτούλαβο, αλλά θα πρέπει να, κάνουμε, να λάβουμε δράση. Συγκεκριμένο τρόπο επιτόπου, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τα κράτη-μέλη για τα θεσμικά όργανα, για τους εταίρους μας, να τους προστατεύσουμε και να ασχέσουμε αυτές τις απειλές πιο αποτελεσματικά. Απαιτείται λοιπόν περισσότερη συνεργασία μεταξύ θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών. Γι' αυτό σας λέω ότι οι περισσότερες απαντήσεις πρέπει να έρθουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό σας είπα ότι μέσα στην οδηγία που αναφέραμε υπάρχουν οι απαντήσεις. Ήδη οι προσπάθειες έχουν αρχίσει και συνεχίζονται. Οπότε η Γενική Διεύθυνση για τα εσωτερικά θα παίξει σημαντικό ρόλο. Και άλλο δυνατό σημείο μας είναι η διαφθορά. Μπορεί να είναι συγκεκριμένες περιπτώσεις, ας πούμε χρηματοδότηση κομμάτων, και αυτό είναι όμως ευάλωτο σημείο. Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να μας απασχολήσουν και αυτή η ομάδα εργασία θα αρχίσει να δουλεύει και έχουμε επίσης τώρα κάποιους πιλότους για αυτό το Fusion Cell που κάνει το εξής μαζεύει πληροφορίες αυτή η ομάδα και αν υποψιαστούν ότι υπάρχουν κριτικές δραστηριότητε επιλήψιμε, αξιολογούν τις, ε, την κατάσταση βάση των πληροφοριών και επί τη βάση αυτής της αξιολόγησης ε, εμείς διατυπώνουμε συστάσεις. Και μετά οι απόκειτες ακρατημέλη να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν με αυτές τις συστάσεις. Τώρα για αυτές τις προτάσεις μας που πρέπει να εφαρμοστούν, αυτό είναι το κρίσιμο σημείο για όλη αυτή τη διαδρομή. Θα είναι ανοιχτό αυτός ο κατάλογος, γιατί πάντω θα επιδέχεται συμπλήρωση και μετά το τέλο του χρόνου, αλλά είπαμε ότι έχουν προτάσεις όπως από τι κάτω χώρε. Ε, θα θα πόσοι κατά την Ολλανδική Προεδρία τις προτάσεις και άλλα κρατημέλια τα οποία θέλουν κοινή δράση ΕΕ ΝΑΤΟ για να αναπτύξουμε αυτή μας την ανθεκτικότητα σε διάφορους τομείς. Οπότε και θα γίνουν συγκεκριμένα διαβήματα, συγκεκριμένα βήματα για να μπορούμε να δημιουργήσουμε τις δυνατότητες και να είμαστε πιο ανθεκτικοί. Είπαμε για τους ε, συμβούλους, για τα υπάρχοντα εργαλεία, ή άλλα. Όλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τελευταίο είναι ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τα κράτη-μέλη να βοηθήσουν αυτή τη διαδικασία. Οπότε συνεχίζουμε επομένω τις κρούσεις στα θεσμικά όργανα. Και μετά τον μπαλάκι θα είναι στο κύπρο των κρατών μελών. Το τι να κάνουν με αυτές μας τις προτάσεις. Πώς θα τις χρησιμοποιήσουν. Τώρα κάτι για ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική ευκαιρία που δεν θα πρέπει να χαθεί. Εάν δεν μπορούμε να βοηθήσουμε για αυτές τις κριτικές απειλές τη συνεργασία Ένωσης ΝΑΤΟ, ε, τότε πότε θα γίνει αυτή η συνεργασία, γιατί είναι τόσο, τόσο χτυπητό, τόσο προφανές ότι έτσι πρέπει να γίνει. Αυτό είναι μέσω πολιτική των κρατών μελών. βεβαίω και τα κράτη-μέλη θέλουν ε, να υπάρχει συντονισμό, συνεννόηση μεταξύ αυτών των εργαλείων, δηλαδή ΕΕ και ΝΑΤΟ. Άρα είναι ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Και σε σχέση με όλα αυτά τα οποία είπε ο Τίμο, να προσθέσω τα εξή δύο. Πολύ σημαντικά. συγχρονισμός στη διαχείριση της κρίσης όταν μια χώρα πλήσεται πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ό,τι μέσο υπάρχει διμερές, πολυμερές θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει την κατάσταση. Και θα πρέπει αυτό να γίνει ταχαίως και με συντονισμό. πρόκειται για τους μηχανισμούς αντιμετώπιση τη κρίση που θα πρέπει να βελτιωθούν, να έχουν συντονισμό και έτσι θα μπορούμε καλύτερα να βοηθήσουμε. Πολύ σημαντικό. Κάτι άλλο τώρα. Εκπαίδευση, ασκήσεις. Και όσον αφορά αυτή την εκπαίδευση, τι θέλουμε να πούμε. Πρώτα-πρώτα είναι το να εκπαιδεύσει κανείς αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. το πώς επίσης μέσω των ε, σχολείων του τόπου της δουλειάς ο κόσμος θα γίνει συνειδητοποιημένος. Γιατί υπάρχουν κάποιοι κανόνες που θα πρέπει να τηρηθούν. Και έτσι θα τα καταφέρουμε να είμαστε πιο ανθεκτικοί. Πληροφορική και άλλοι τομείς που πρέπει να επισημαθούν. Εδώ θα βάλω τελεία. Δεν υπάρχει πρόβλημα κύριε Διευθυντά και σας ευχαριστούμε για αυτήν την πλήρη και τόσο ενδιαφέρουσα ομιλία σας. Και τώρα, ο κύριος Ρικ Βάιλες, ο οποίος εκπροσωπεί την Λετωνία. Εκεί υπάρχει συνειδητοποίηση του ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί αντοχή κατά του υβριδικού πολέμου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Φωτίδη. Άκουσα τι ελέγχθη. Και ελέγχθησαν πολλά. Οπότε, για να δούμε τι απομένει να πει κάποιος εκπρόσωπος μιας εθνικής κυβέρνησης. Συμφωνώ κύριε με αυτά τα οποία είπατε. Άρα να μην επαναλάβω το πόσο παλιά υπόθεση είναι οι υβριδικές τακτικές, οι υβριδικοί πόλεμοι. Οπότε η γνώση της αντιμετώπισης τους, αυτών των φαινομένων, αυτών των πολέμων, επίσης είναι παλιά στα θεσμικά όργανα. Ήδη από το 57 Θεωρείται ότι το να υπάρχει αποτροπή πυρηνική από κάποια συμμαχία, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποιες επιχειρήσεις. Επιλέξει, λέγανε, με περιορισμένους στόχους όπως διείσδυση ή κάποιες ε, ε, επιθέσεις στην περιοχή ε, ευθύνη του ΝΑΤΟ. Οπότε οι σύμμαχοι έτσι θα μπορούσαν να περιορίσουν τη δράση, θα μπορούσαν να περιορίσουν τη δυνατότητα πολέμου ή θα μπορούσαν να διαλέξουν να μην αντιδράσουν καθόλου. Αυτό είχαν τότε επιλέξει. Οπότε υπήρχε αυτή η έννοια, αυτή η σύλληψη του τι είναι εχθρός και πώς μπορεί να τον παραλύσει κανείς. Είναι κάτι παλιό επομένως στην αντίληψή μας για την ασφάλεια και αυτό το δόγμα αναπτύχθηκε περισσότερο το 68 όσον αφορά την άμυνα και τη στρατηγική, όσον αφορά τα εργαλεία λήψη αποφάσεων, ούτω ώστε να μπορεί κανείς να λάβει ταχύως αποφάσεις. Πάρα πολλά από αυτά τα στοιχεία που οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν υπήρχαν από παλιά και η γνώση του προβλήματος. Επομένως είναι καλά μαντάτα αυτά για τη χώρα μου. Το ότι υπάρχει κατανόηση ε, αυτών των ε, θεμάτων και ότι αυτά βγήκαν από το χρονοτούλαπο και επανήλθαν στην επικαιρότητα. Βέβαια τα πράγματα και οι συνθήκες έχουν κάπως αλλάξει από τότε. Κρίμα όμως που αναλάβαμε δράση μόνο όταν στριμωχτήκαμε. Γιατί το 2011 ήδη τον προσπάθησε να αντιμετωπίσει αυτές τις ε, υβριδικές απειλές. Και γίνανε σχετικές κινήσεις, αλλά τέλος πάντων δεν προχώρησε αρκετά και έτσι κατά κάποιο τρόπο χάθηκαν τρία χρόνια. Προφανώς και το ότι ο επιτιθέμενος, ο εχθρός, θα έχει συνδυασμό στοιχείων που θα χρησιμοποιήσει, δεν μπορούμε να το προβλέψουμε ακριβώ όλα. Οπότε θα πρέπει να προσέξουμε να μην ε, εθελοτυφλούμε. Δεν θα είναι το σκηνικό ξεκάθαρο σε περίπτωση απειλής. Άρα, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες ε, απειλέ και να τι καταπολεμήσουμε όποτε χρειάζεται θα πρέπει μια κυβέρνηση να συνδυάσει διαφορετικές μεταβλητές και δυνατότητες. Βούληση και όχι μόνο πολιτική λήψη αποφάσεων, βούληση της κοινωνίας για αντίσταση. Για να σας πω τι εννοώ με, αυτέ, με αυτές τις έννοιες, αυτές τις μεταβλητές. Για τις δυνατότητες, όπως ακούσα τους προλαλήσαντες, ε, αυτό το θέμα είναι ευρύτατο. Πού να τα καλύψουμε όλα. Πού να καλύψουμε όλα μας τα μειονεκτήματα και δύνατα σημεία. Αλλά χρειάζεται να υπάρχει συνέστηση, συνειδητοποίηση της γενικότερης κατάστασης και επίσης να υπάρχει επαρκής ε, ε, λήψη πληροφοριών. Γιατί πολλές φορές έχουμε πληροφορίες, αλλά υπάρχουν προβλήματα. Προβλήματα δηλαδή ότι το ένα θεσμικό όργανο δεν μπορεί να τα πει στο άλλο, το ένα κράτος στο άλλο και οπότε έτσι, όπως αναφέρθηκε, θα πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός εκ των προτέρων και επίσης να υπάρχει επαρκής μηχανισμός προειδοποίησης. Ιδίως όσον αφορά την προστασία των συνόρων. Όπως διαπιστώθηκε, το θέμα της ασφάλειας των συνόρων δεν είναι εύκολο. Δεν είναι απλό. Και από τα, τι θα γίνει στα σύνορα εξαρτάται τι θα γίνει στην ενδοχώρα. Άρα θα πρέπει κανείς να μπορεί να είναι αποφασιστικός κατά του εισβολή. Αυτό βέβαια προϋποθέτει υλικό, αμυντικό και εκπαίδευση των μονάδων, των, των ανθρωπίνων πόρων. Άρα θα πρέπει να εμπλεκούν οι τοπικές αρχές ασφαλείας αλλά και οι εθνικές αρχές ασφαλείας καθώς και επίσης να κινητοποιηθούν και οι συμμαχικές δυνάμεις μεταξύ κρατών μελών. Άρα χρειάζεται κινητοποίηση, δυνατότητα κινητοποίηση τέλο πάντων. Και να υπάρχει συντονισμό όταν έρθουν να βοηθήσουν οι σύμμαχοι. Οπότε θα πρέπει να προετοιμαστούμε για μακρά περίοδο συγκρούσεων, αλλά και για υψηλή ένταση αυτών των συγκρούσεων. Τέτοια ε, διαδικασία να ε, ληφθεί υπόψη. Άρα χρειάζεται να υπάρχει η κρίσιμη υποδομή. Αυτό αφορά και το ηθικό, αλλά και την έρευνα όπως αναφέρθηκε. Χρειάζεται να υπάρχει αυτό που λέμε ανωτερότητα στην πληροφόρηση από πλευρά της συμμαχίας. Αυτό αφορά τα αφηγήματα, αυτό αφορά τα μηνύματα επίσης τα οποία στέλνουμε. Και θα πρέπει να αναπτύξουμε μια ούτως πειν ιατροδικαστική της εισβολής για να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. αυτά τα πράσινα ανθρωπάκια που λένε, αυτοί οι κομμάντος δηλαδή, οι, αυτές οι πολιτοφυλακές, από πού προέρχονται. Και να μπορούμε όλα αυτά να τα προβάλλουμε και να τα αποδείξουμε στους συμμάχους μας. Γιατί το πρόβλημα το τι γίνεται όταν δύο ομάδες ε, εθνών πρέπει να συνοηθούν, το πρόβλημα είναι ότι οι μένου ρωτούν τους δε πώς μπορείτε να αποδείξετε ότι γίνονται τέτοια πράγματα από πού και ως πού αυτές οι δυνάμεις ανήκουν στο τάδε κράτος. Άρα, γι' αυτό πρέπει να υπάρχει αυτή η ιατροδικαστική ούτως υπήν δυνατότητα απόδειξης. Ετοιμότητα, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα πρέπει να υπαρχει αυτη η ιατροδικαστικη ουτως δυνατοτητα αποδειξης ετοιμοτητα που ειναι παρα πολυ σοβαρο θα πρεπει να υπαρξει σε όλες χώρες για την εθνική ασφάλεια. Αυτή είναι η δουλειά και το καθήκον θα πρέπει να έχουμε. Και αυτό καλύπτει και τον κρατικό κορβανά, εκπαίδευση αστυνομίας, παραστρατιωτικούς, ειδικέ δυνάμεις, υποδομή και αλλαγή νοοτροπίας. Άλλο τώρα. Αλλη... Διαδικασία λήψη αποφάσεων. Όταν λοιπόν κάποιο είδου εισβολή και υβριδικές τακτικές τότε θα πρέπει να υπάρχει έγκαιρη, γρήγορη λήψη αποφάσεων. Πολύ σημαντικό αυτό. Συγχρονισμός σε επίπεδο κράτους. Να συνειδητοποιηθεί ότι το κράτος είναι ο πρώτος αποδέκτης τέτοιων ενεργειών και για τον ΝΑΤΟ ισχύει αυτό, όπου βέβαια έχουμε το θέμα της συλλογική απόφαση. Επίσης, πολλές φορές έχουμε λήψη αποφάσεων μόνο από κάποιους αξιωματούχους. Βεβαίως ε, υπάρχουν θέματα όταν το πολίτευμα είναι δημοκρατικό, αλλά να μην θεωρούμε ότι λόγω αυτού είμαστε σε κατώτερη θέση. Γιατί βεβαίως και οι αποφάσεις λαμβάνονται επί τη βάση πληροφοριών και υπάρχει σχέση μεταξύ κατασκοπίας πληροφοριών και μειονεξίας ε, αδύνατων σημείων σε σχέση με την επισήμανση της απειλής. Άρα θα πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση, θα πρέπει να είναι κάποιος εξασκημένος. Και αυτό θα πρέπει να γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Πολύ σημαντικό. Σε όλη την πυραμίδα από τους ηγέτες μέχρι τους, ε, τους κομμάντους αυτούς οι οποίοι δρούν στη, βάση της πυραμίδας. Να ξέρει δηλαδή ο καθένας τι πρέπει να κάνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Όχι, όχι ο καθένας να κάνει το κεφαλίου του ε, και να μπορεί να δράσει αυτόνομα, που και αυτό είναι σημαντικό, αλλά να ξέρουν τις διαδικασίες, να ξέρουν τις αρμοδιότητες και ευθύνες και να ξέρουν πώς θα το κάνουν από πλευράς χρόνου και χώρου. Άρα, λήψη αποφάσεων που επιδέχεται και αυτή η εκπαίδευση, ακόμα και σε αυτές τις θολές καταστάσεις, τους θολούς αυτούς πολέμους, Οπότε έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα μπορέσουν να μπορούν να αντιδράσουν καλύτερα και συλλογικά. Όσον αφορά τώρα τη βούληση ανταπόκρισης και αντίστασης ε, αυτό είναι θέμα που πάει και παραπέρα από το θέμα συμμαχίας, από το θέμα επιρροής Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σε επίπεδο εθνικό αυτό είναι θέμα της στρατηγικής ελίτ και της κοινωνίας, να εξασφαλίσουν το πώς θα διαδοθούν, πώς θα πιάσουν ρίζες ή κάποιες αξίες που έχει κάθε χώρα. Και εδώ είναι απαραίτητο να υπάρχει ηγεσία για να ληφθούν κάποιες σημαντικές αποφάσεις και να υπάρχει ηγεσία την ώρα της κρίσης. Αυτό μπορεί να μην είναι σύμφυτο με την στρατηγική και να το βρίσκει κανένας όποτε θέλει, αλλά σίγουρα χρειάζεται. Για κυβερνόπηλες επομένως, εκτός από την προετοιμασία κάποιου κράτους, τι άλλο μπορεί να γίνει η χώρα μου πάντα πίστευε ότι και η Ένωση και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να δρουν ε, σε συνεργασία και συμπληρωματικά. Οπότε αυτά τα οποία γίνονται τώρα, ακριβώ αυτά που είπαν οι συνάδελφοι εκ δεξιών μου, όλα αυτά τα χαιρετίζουμε, τα θεωρούμε πολύ θετικά ως χώρα. Και θα πρέπει να διευκολυνθούν οι σχετικές δράσεις όσο γίνεται περισσότερο γιατί θεωρούμε ότι κάθε υβριδική κρίση μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με συμπληρωματικότητα αυτών των δύο φορέων ε, και και το και βάλαμε ικανοποίησή μας ακούσαμε ότι υπάρχουν διαδικασίες και κινήσεις πολύ επικοδομητικό αυτό και συμφωνώ ότι δεν πρέπει να κολλάμε τώρα στον τον ορισμό τη έννοια υβριδικό. Αυτό δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Αυτό τους υβριδικές, ο υβριδικό πόλεμο είναι κάτι σαν ένα ιό που μεταλλάσσεται, να, το 40 η Λετωνία αντιμετώπισε τέτοιε υβριδικέ απειλές και επιχειρήσεις από την Σοβιετική Ένωση. Αλλά αυτό δεν είναι αναγκαστικά το ίδιο με τι έγινε το 1978 στο Αφγανιστάν, ούτε με τι έγινε το 2014 στην Ουκρανία ή τι γίνεται τώρα, τώρα ή τι θα γίνει σε ό,τι τυχόν συμβεί στο μέλλον. Νομίζω πολλές απειλές η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουμε και πολλά μέσα αντιμετώπιση στη διάθεσή μας. Ούτε το ΝΑΤΟ ε, ενίσταται σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει αυτές τις βρετικές απειλές και να χτίσει αντοχή. Ε, επίσης, να ληφθεί υπόψη ότι αυτές οι απειλές μπορεί να έχουν και πυρηνική πτυχή και συμβατική. Και αυτό είναι θέμα του ΝΑΤΟ βασικά. Άρα έχει τεράστια σημασία η συνεργασία Ένωσης ΝΑΤΟ. Εν κατακλείδη για να δούμε κάποιους, ε, κάποιους μεταβλητές που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικέ. Θα πρέπει να έχουν συνεπή δράση και οι δύο φορείς. Η στρατηγική του ΝΑΤΟ. Αυτά που είπε ο Αμπλωτής Γενικός του ΝΑΤΟ πρόσφατα. σε κάποιο σεμινάριο για το πώς κανείς να προετοιμάσει την αμυνά του, την αποτρεπτική. Και είπε ότι και η Ένωση για το να τον μπορούν να εξασφαλίσουν ανάπτυξη άμυνας και θα πρέπει βέβαια να κατανοήσουμε καλύτερα τι θα πει αποτροπή. Διότι αποτροπή δεν πάνε να πει μόνο στρατιωτική δράση, στρατιωτική αντίληψη. Έχει πολύ σημαντική πτυχή, οικονομική, πολιτική, και άλλες πτυχές. Όποιοι ασχολείστε με αυτόν τον τομέα, ε, ξέρετε πόσο ευρεία είναι η έννοια της αποτροπής. Δηλαδή χρειάζεται να καταλάβει ο εχθρός ότι εάν επιτεθεί αυτό θα του κοστίσει ακριβά. Όμως αποτροπή σημαίνει επίσης και την παρουσία συμμεχικών δυνάμεων στην επικράτεια κάποιου κράτους. Και αυτό στέλνει μήνυμα αποτροπής ηχηρό. Ε, επίσης αναβάθμιση των ε, μυντικών δυνατοτήτων να μην ε, υπάρχουν ασάφειες στη διαχείριση αυτών των μέσων, αλλά βέβαια δεν μπορεί κανείς να προτείνει κάτι που να ισχύει για όλους, γιατί κάθε χώρα είναι διαφορετική, επομένως θα πρέπει να γίνεται περιπτωσιολογική, εξατομικευμένη προσέγγιση και να βλέπουμε τα δυνατά σημεία του, του κάθε κράτους ε, χωριστά τη συνεργασία με τους συναδέλφους ΕΝΑΤΟ και Ένωση. Ε, μια τρίτη αρχή σημαντική θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και με την ενίσχυση σε περίπτωση επίθεση. Και δεν εννοώ μόνο από πλευρά στρατιωτική. Δεν λέω ότι αυτό είναι εργαλείο μόνο στρατιωτική φύσεω. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες ειδικέ δυνάμεις, ειδικέ μάλλον επιχειρήσεις ακόμα και από την αστυνομία σε περίπτωση κυβερνοαπειλής και να υπάρχει στρατηγικό υλικό ε, ή σε επίπεδο ενέργειας να υπάρχουν κάποια μέσα ε, τα οποία να χρειάζονται αντίσταση γιατί όταν κόβονται οι πόροι από κάποια χώρα ε, τότε αργά ή γρήγορα η σε επιπεδο ενεργειας να υπαρχουν καποια μεσα τα οποια να χρειαζονται αντισταση γιατι οταν κοβονται οι ποροι απο καποια χωρα τοτε αργα η γρηγορα η χωρα δεν θα μπορεί να αμυνθεί σε κάποια απειλή. Τέλος δε, να επανέλθουμε στο πόσο σημαντικό είναι το να υπάρχει ενότητα προσπαθειών όσον αφορά την επικοινωνία. Τα αφηγήματα να συνεχίζουν να προβάλλονται και να γίνονται κατανοητά. Δηλαδή, να λέμε ότι λέμε, να το λέμε ξεκάθαρα. Όπου και να τα λέμε, να το ακούνε. Και κυρίως να παρατεθούμε στην εχθρική προπαγάνδα. Οπότε γι' αυτό και σας λέω, εάν μπορούμε να έχουν προσπάθειες επιτυχής, συντονισμένες, να ισχύσουν οι αποφάσεις ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, να υπάρχει συνεργασία των ε, πρωτευουσών, τότε θα ε, βρεθούμε νικητές στο παιχνίδι αυτό έναντι των αντιπάλων. και να λέμε υπόψη πάντα την ιδιωτική κατάσταση γιατί όλα αυτά δεν έχουν παγκόσμια ισχύ για όλους. Σας κατευχαριστούμε. Και οι τρεις παρουσιάσεις ήταν τόσο πλήρεις που τα πολυπληθή μέλη εδώ είναι πολύ ικανοποιημένα Όμως η κυρία Λόζινγκ θέλει το λόγο παρόλα αυτά. Θα μιλήσω στα γερμανικά, αλλά κυρία Λόζινγκ, βάλτε τα ακουστικά σας και θα περιμένω λίγο. Και σας ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα κατά την άφηξή μου και δυστυχώς ε, είχα και άλλες υποχρεώσεις πριν την συνεδρίαση της Επιτροπής. Ενδεχομένως λοιπόν να ρωτήσω πράγματα τα οποία ήδη έχετε αναφέρει Ελπίζω πως δεν θα κάνω ερωτήσεις που, δεν έχουν, που έχουν ήδη απαντηθεί. Είπατε στο τέλος ότι θα πρέπει να μην εστιάσουμε τόσο πολύ στον ορισμό των ευρετικών ε, απειλών. Το καταλαβαίνω αυτό. Και ακούγοντας από τον κύριο Κλόντι ότι προωθούνται συγκεκριμένα μέτρα Είναι αντίθετο με την ε, ασαφή αυτή έννοια που αναφέραμε προηγουμένως. Και πιστεύω ότι είναι κάπως προβληματικό αυτό. Και δεν είμαι και η μόνη που θεωρεί ότι είναι προβληματικό αυτό. Έχουμε και ένα άρθρο από την αναθεώρηση του ΝΑΤΟ για τους εμπρετικούς πολέμους, κατά πόσον υπάρχουν καν. Από τον ορισμό φυσικά προκύπτουν και τα μέτρα. Αναρωτιέμαι λοιπόν κατά πόσον σε αυτό το ασαφές πλαίσιο οι διαφορετικοί παράγοντες όπως το Ισλαμικό κράτος, η Ρωσία ή διαφορετικά φαινόμενα όπως, διάφορα φαινόμενα όπως η οργανωμένη κλιματικότητα, η χρήση ειδικών μονάδων χρησιμοποιούνται μεν, αλλά σε ένα σαφές πλαίσιο. Αυτό σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να το συζητήσουμε. Μήπως ο όρος αυτός είναι και θα παραμείνει υπερβολικά σαφής; Φυσικά, σε θέματα περιγραφής μέτρων ασφαλώς και θα συγκεκριμενοποιηθεί. Η κυρία Μογκερίνη στο έγγραφο Food for Thought περιέγραψε με ακρίβεια τι μέτρα χρησιμοποιήθηκαν, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά Ρωσία. Μέτρα και παραθέτω ότι ο παράγοντας επίθεσης μπορούσε να ενισχύσει τα στρατεύματά του. Αυτά τα βλέπουμε λοιπόν ότι γίνονται και από πλευρά της Δύσης στη Συρία, για παράδειγμα. Και φυσικά αυτό έχει συνέπειε. Δεν θέλουμε να κατηγορούμε μεν τους δε. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Αλλά θα ήθελα να θέσω και τους κινδύνους των υβραδικών αυτών απειλών για αυτούς που τις εφαρμόζουν. Για παράδειγμα, για τη Δύση όταν ε, συντάσσει κανείς ε, και αναβαθμίζει τα στρατεύματά του, μετά δεν μπορεί να τα ξεφορτωθεί έτσι εύκολα. Άρα πιστεύω ότι ενέχονται κίνδυνοι όχι μόνο από το ότι δεν ξέρουμε το πώς θα δράσουμε, αλλά και από το ότι οι δράσεις αυτές μπορεί να αποβούν πολύ επικίνδυνες. Γι' αυτό λοιπόν θα, θα ήθελα να τονίσω ότι θα πρέπει να υπάρχει πιο συγκεκριμένη περίληψη και συμπερίληψη των κινδύνων και να σκεφτούμε και τις συνέπειες των μέσων βραχυπρόθεσμα, πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Γιάννου Ζεύκαμπ. Εάν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πάρω το λόγο και να μιλήσω ε, και να ευχαριστήσω του προσκεκλημένους μας. Να σας ευχαριστήσω και εσάς για το γεγονός ότι βάλατε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής μας. Τώρα πρέπει να δούμε πώς θα μαζευτούν όσο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και πώς θα γίνει ανταλλαγή απόψεων και σκέψεων για τα φαινόμενα αυτά. Θα ήθελα να συνεχίσω από αυτόν που είπε η κυρία Λούζινγκ. Είπατε κυρία μου ότι όλα αυτά είναι ασαφή λέει εγώ θα σας απαντούσα ότι αυτό ακριβώς είναι το θέμα του υβριδικού πολέμου. Οι υβριδικές απειλές σε αυτό βασίζονται, σε αυτό το ακαθόριστο, απροσδιόριστο στοιχείο. Έτσι έλεγε και ο Κλάουζεβιτς, για να καταλάβει κανείς ένα κράτος πρέπει να εισβάλλει στο, στην επικράτειά του. Αυτό δεν ισχύει όμως τώρα πια. Υπάρχουν καταστάσεις στο σύγχρονο κόσμο όπου υπάρχει σύραξη δύο στρατών όλο και σπανιότερα. Υπάρχει ακόμα, αλλά σπανίζει πια. Τώρα διάφοροι παράγοντες και τα κράτη με άλλο τρόπο θέλουν να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους. Δεν χρειάζεται πολύ συγκεκριμένος ορισμός του υβριδικού πολέμου, αλλά γενικότερα να δούμε περί τίνος πρόκειται. Είναι συνδυασμός πολλών στοιχείων και η πρόσφατη εμπειρία δείχνει ότι αυτές οι απειλές χρησιμοποιούν μη στρατιωτικές μεθόδους όλο και περισσότερο αυτό φάνηκε από τις κυβερνοεπιθέσεις κλπ. Όλη αυτή λοιπόν η συζήτηση για τον υβριδικό πόλεμο και τις υβριδικές απειλές είναι πολύ σημαντικές γιατί αν δούμε μόνο τις στρατιωτικές απειλές τότε βλέπουμε ότι αυτές δεν είναι οι πιο επικίνδυνες. Αντίθετα άλλου είδους απειλές επίκυνται και τις βλέπουμε κάθε μέρα και είναι πραγματικότατες. Θα έλεγα μάλιστα ότι αυτού του είδους οι υβριδικές απειλές δεν είναι απλώς πραγματικές, αλλά είναι και αυξανόμενες. Μπορούμε να αναμένουμε ότι στο μέλλον θα υπάρχουν μόνο τέτοιου είδους απειλές. Αυτές είναι οι κύριες απειλές σήμερα. Κατ' εμέ λοιπόν ένα ιδιαίτερο στοιχείο υβριδικής απειλής είναι η εξής να επιτευχθούν οι στόχοι εξ αποστάσεως, εκ μεγάλης μάλιστα αποστάσεως. Αυτό δεν το αναφέρατε τη γεωγραφική απόσταση. Χιλιάδες χιλιάδων χιλιόμετρων από την Ευρώπη, από ένα γραφείο, από μια επιχειρησιούλα των μυστικών υπηρεσιών, μπορεί κανείς από πολύ μακριά επαναλαμβάνω να απειλήσει την Ευρώπη. Κατ' εμέ υπάρχουν τρεις τομείς που αφορούν ιδιαίτερα την Ευρώπη όπου είναι πολύ ευάλωτη. Πρώτον η προπαγάνδα, ο πόλεμος των νοοτροπιών. Και πρέπει να σας πω ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ αδύναμη να, για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους προπαγανδιστικές απειλές. Και γιατί είμαστε τόσο ευάλωτοι, διότι οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι αυτά τα θέματα δεν πρέπει να συζητιούνται καν κλπ. Δεύτερο αδύνατο σημείο. Η ενέργεια Χωρίς την ενέργεια δεν μπορούμε να κρατήσουμε τον πολιτισμό μας. Και τρίτο αδύνατο σημείο η πληροφορική, το νέο είδος επικοινωνίας. Πριν έπρεπε κανείς να βομβαρδίσει αεροδρόμια, τώρα αρκεί να καταστρέψει τα πληροφορικά συστήματα ενός αεροδρομίου από μεγάλη απόσταση. Το είδαμε και στο Ζάβιντεμ. Όλο το αεροδρόμιο παρέλυσε πολλές ώρες και δεν ξέρουμε ακόμα γιατί. Εδώ λοιπόν βρίσκονται οι μεγάλες απειλές. Και εδώ πρέπει να δράσουμε και να αντιδράσουμε για να τις αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, εγώ έχω ακόμη αμφιβολίες ως προς την αποτελεσματικότητα του συντονισμού των ευρωπαϊκών δράσεων και επιχειρήσεων. Και από εσά, από ό,τι είπατε κύριε, φάνηκε αυτό ότι υπάρχουν προσπάθειες αντίδρασης και εμείς αναμένουμε πάντοτε από τα κράτη που υφίστανται επίθεση να αντιδράσουν πρώτα. Ναι, αλλά αν υπάρξει επίθεση ταυτόχρονη κυβερνοεπίθεση ή του, κατά του τραπεζικού συστήματος πολλών κρατών ταυτόχρονα εφόσον μάλιστα και οι τράπεζες είναι όλες μεταξύ τους συνδεδεμένες τότε τι γίνεται έπειτα τα κράτη έχουν πολύ διαφορετικές δυνατότητες αντιμετώπισης τέτοιων απειλών μερικά δεν κάνουν τίποτα δεν μπορούν να αμυνθούν. Ερωτώ λοιπόν, έχετε αναλύσεις αποτελεσματικότητας των διαφόρων κρατών για την αντιμετώπιση τέτοιων απειλών και αν έχετε τέτοιες αναλύσεις ετοιμότητας και δυνατότητας μήπως θα έπρεπε να σας πω μάλλον ότι η Ολλανδία θαύμασα γιατί μπόρεσε να αντιμετωπίσει μια τέτοια κυβερνοεπίθεση πράγμα που δεν ήταν και πολύ εύκολο. Σας ευχαριστώ κύριε μου, κύριος Μπούχνερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, παρουσιάσεις σας και με... Ε, πραγματικά είμαι πολύ ικανοποιημένο ε, που το οργανώσαμε αυτό το θέμα. Θα ήθελα να αναφερθώ στις εσωτερικές αναταραχές. Μπορεί να υπάρχουν λοιπόν εξωτερικές επιθέσεις ή ενδεχομένω ε, τέτοιες εσωτερικές ανησυχίες μπορούν να δημιουργηθούν αυτόνομα αλλά να τις εκμεταλλευτούν εξωτερικές δυνάμεις. Αυτό σίγουρα το έχετε λάβει υπόψη. Είπατε ότι είναι δύσκολο να συντονιστούν οι μυστικές υπηρεσίες των διαφορών κρατών μελών και να υπάρξει ανταλλαγή τέτοιων ε, πληροφοριών. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πολύ συγκεκριμένα ποια είναι εδώ πέρα, ποιος είναι ο ρόλος των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς αντιδρούμε σε τέτοιες ε, περιπτώσεις έναντι τέτοιων απειλών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρος. Και τώρα θα ήθελα να παρουσιάσω και εγώ δύο ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με την στρατηγική επικοινωνία Stratcom στο πλαίσιο του υβριδικού πολέμου. Νομίζω ότι βάσει των συζητήσεών μας ε, των τελευταίων χρόνων συνειδητοποιούμε τις απειλές που προέρχονται εξ Ανατολάς. πριν την προσάρτηση της Κρυμαίας κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και αυτό βασικά προέρχεται από το κέντρο αριστείας ε, με βάση, τη, με βάση τη Ρήγα που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής ΣΕΝΤΕ. Ξέρουμε ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαΐου ήταν αυτά που ήταν και τα περαιτέρω πορίσματα του Συμβουλίου του Ιουνίου. Ξέρουμε ότι εισήγαγαν κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση των δράσεων αυτών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. αλλά υπάρχουν και αναφορές για εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί από το Days. Πείτε μας, έχει αναλυφθεί οποιαδήποτε δράση για να γίνει συντονισμός και να μοιραστεί, κατανεμηθεί αυτή η γνώση. Κατά δεύτερον, υπάρχουν νέες εξελίξεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα τεράστιο κύμα μετανάστευσης. Ποιος είναι ο αντίκτυπος σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα. Τι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Τι θα πρέπει να κάνουμε. Προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά μας. Σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς. Να δώσω το λόγο τώρα στους πανελίστες με την ίδια σειρά που μας ε, έκαναν την παρουσίασή τους, ενδεχομένω να υπάρξει και δεύτερο γύρος. Έχουμε μείνει λίγο πίσω, αλλά θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε λίγο αυτοσυγκράτηση στο χρονομιλές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, δεν θα μακρηγορήσω. Θα ήθελα να θέσω το θέμα στο οποίο αναφέρθηκε η κυρία Λούζινγκ. Είναι πρόβλημα άρα για το γεγονό ότι, ότι δεν υπάρχει ορισμός επί του οποίου έχουμε συμφωνήσει και αν δεν υπάρχει ορισμός πώς μπορούμε να δούμε ποιες είναι οι δράσεις που απαιτούνται. Να επανέλθω σε κάτι που υπάρχει. Δεν υπάρχουν δύο παρόμοια υβριδικά σενάρια. Από τη στιγμή λοιπόν που θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε κάτι, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα στην επόμενη βρετική επίθεση. Εμείς προσπαθούμε να εντοπίσουμε τους συντελεστές που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογή των βρετικών πολέμων που ενδεχομένως να αλλάξουν στη σύνθεσή τους, στο συνδυασμό τους. Δεν είναι πολύ πιθανό να έχουμε μικρά πράσινα ανθρωπάκια στο επόμενο υβριδικά, σε επόμενε ευρυδικέ απειλέ. Μπορεί το επόμενο σενάριο να είναι διαφορετικό, καταλαβαίνετε. Εντελώς διαφορετικό. Προσπαθήσαμε λοιπόν να εντοπίσουμε τουλάχιστον ποιο είναι το πεδίο, το εύρος, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει μια τέτοια επίθεση. DIM, e, DIM e διπλωματικές πληροφορίες για στρατιωτικές, οικονομικές και μυστικές και νομικές πληροφορίες. Όλοι αυτοί οι τομείς λοιπόν. Μπορούν να περιληφθούν και μπορούν να περιληφθούν και να εμφανιστούν επί τόπου. Αλλά μπορεί να παρουσιαστούν και εκτός της επικράτειας μας συγκεκαλυμμένα ή και εμφανώς. Κάποια εξ, αυτών δεν είναι καν παράνομα. Δεν είναι παράνομο, για παράδειγμα, να ασκηθεί προπαγάνδα. Δεν είναι παράνομο να συσταθεί μία μικιό σε μία άλλη χώρα. Δεν είναι εξορισμού ε, για παράδειγμα παράνομο, να εκδοθούν ρωσικά διαβατήρια για τη ρωσική μειονότητα στην Κρυμαία. Απλά εμείς αυτό που εντοπίζουμε είναι τους παράγοντες, τους δείκτες, τους συντελεστές που μας επιτρέπουν να πούμε ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Κάτι έκτακτο, εξαιρετικό, στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας. Κοινωνική αναταραχή. Η κοινωνική ανταραχή από μόνο της δεν αποτελεί ένδειξη βρετική επίθεση. Σε αυτή την πόλη, για παράδειγμα, έχουμε εδώ πολλέ κοινωνικέ ανταραχέ. Έχουμε διάφορε εκπρο... διάφορες ομάδε εκπροσωπήσει πολιτών, αντιπροσωπήσει πολιτών που έρχονται να διαδηλώσουν εδώ στι Βρυξέλλε. Αυτό από μόνο του δεν αποτελεί ένδειξη βρυδική απειλή. Πρέπει λοιπόν να καταλαβαίνουμε καλύτερα τι συμβαίνει και να μπορέσουμε να συνδέσουμε αν θέλετε τις τελίτσες για να δημιουργηθεί μια εικόνα και να αποφασίσουμε τελικά αν πρόκειται για κάτι το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά κανονικών γεγονότων, φαινομένων, τα οποία όμως συνθέτουν την επαρχή μιας ε, υβριδικής επίθεσης. Στο τέλος δεν είναι δύσκολο φυσικά να καταλάβουμε από πού προέρχονται αυτά τα ζητήματα. Αλλά τι γίνεται στην πορεία. Πριν καταλήξουμε στην ε, κανονική στοχευτική σύγκρουση. Αυτό θα πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα. Α, αυτό μπορεί να μην μας ικανοποιήσει κάθε περίπτωση. Μπορεί να μην το εντοπίζουμε πάντα με τον σωστό τρόπο, αλλά αυτό είναι και το δύσκολο. Αυτή είναι και η πρόκληση. Να μπορέσουμε να λαμβάνουμε αποφάσεις σε περιβάλλοντα ασάφειας και αβεβαιότητας. Εντάξει, ναι, άμα δεκάδες χιλιάδες ε, περάσουν τα σύνορα, είναι εύκολο να πούμε ότι πρόκειται για ρωσική επίθεση. Σε ό,τι αφορά την Κρυμαία, το σημείο αυτό της Ουκρανίας. Αλλά αν δεν υπάρχει 100% βεβαιότητα και πάλι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και θα πρέπει παρόλα αυτά να, συ, συλλέξουμε όσο πιο πολλές πληροφορίες γίνεται μεταξύ των οργανώσεων και όχι μόνο μεταξύ ΝΑΤΟ και, ε, και Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΑΣΑ για παράδειγμα έχει πολλούς τοπικούς παρατηρητές που μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τι γίνεται αλλά και μεμονωμένους πολίτες. Πολλές πληροφορίες είναι open source ε, αυτά που βλέπουμε για παράδειγμα στις εφημερίδες, αυτά που παίρνει φωτογραφία ο πολίτης στο δρόμο. Άρα πρέπει να συνενώσουμε και να αναγνωρίσουμε τη φύση όλων αυτών των φαινομένων προκειμένου να λαμβάνουμε αξιόπιστες αποφάσεις. Και αυτό ακριβώς προσπαθούν να αποφύγουν οι εχθροί μας. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ασάφειας και αβεβαιότητας. Είτε πρόκειται για ε, κράτη είτε όχι. Σας ευχαριστώ κύριε Κλοντή. Ωραία. Φυσικά υπάρχει μια τάση χρησιμοποίησης της ονομασίας υβρίδιο για πολλά πράγματα. Οι υβριδικές απειλές ακούγονται πολύ συχνά και είναι της μόδας. για να δοθεί περισσότερη προσοχή σε ό,τι ονομάζεται υβριδική απειλή. Αυτό σίγουρα. Αλλά θα έλεγα ότι αντί για ορισμό, που είναι κάτι πολύ δύσκολο, αυτό που χρειάζεται είναι μια συμφωνία ακόμη και εθνικά. Θα ήταν δύσκολο να οριστεί. πόσο μάλλον από μια ευρύτερη κοινότητα. Πώς να συνδυάσουμε λοιπόν αυτά που έχουμε δει στην Ανατολή, στην Ανατολική Ευρώπη, μπροστά στα μάτια μας, αν μπορούμε δηλαδή να τα ονομάσουμε υβριδική απειλή. Ποιος ξέρει και πόσες άλλες θα δούμε στο μέλλον. Αντί λοιπόν για ορισμό. In the UN, uh, of... Uh, ας πούμε για την τρομοκρατία, ας πούμε για την τρομοκρατία. Αντί λοιπόν για ορισμό που είναι κάτι πολύ δύσκολο και ίσως και αμφιλεγόμενο και δεν εξυπηρετεί και κανένα σκοπό, καλύτερο είναι να υπάρξει μια κατανόηση του τι είναι οι βρυδικές απειλές και συνεχώς να την ενημερώνουμε την περιγραφή αυτή. Δεν είναι φωτογράφηση ότι ό,τι κατανοούμε σήμερα ως βρυδική απειλή θα είναι και σε πέντε χρόνια το ίδιο. Μα οι υβριδικές απειλές ακριβώς συνεχώς αλλάζουν Πρέπει λοιπόν αυτό να το ξέρουμε. Αυτές λοιπόν οι συνεχώς ανανεούμενες και αλλάζουσες καταστάσεις μπορεί να συμπεριλαμβάνουν όλο και περισσότερους τομείς που να μας δείχνουν πού ακριβώς πρέπει να ενδιαφερθούμε. Το θέμα δεν είναι ο ακριβής ορισμός εφόσον καταλάβουμε ότι υπάρχουν απειλές και τροτά σημεία που πρέπει να τα γνωρίζουμε και που απαιτούν κάποια αντίδραση εκ μέρους μας. Αν αυτό γίνει κατανοητό και είναι ο στόχος μας, τότε μπορούμε να τον πετύχουμε. Τώρα σε κάτι που έλεγε ο Τίμος προηγουμένως. Η δοκιμή, η δοκιμή για τα τροτά σημεία και για να τα πούμε με όρος ΝΑΤΟ το να παραμείνουμε κάτω από το άρθρο 5. Πώς μπορεί να υπάρξει αποσταθεροποίηση χωρίς πολύ ομή αντίδραση. Αυτό είναι το άρθρο 5. Ξέρουμε ότι πολλές υβριδικές απειλές μπορούν να καταλήξουν σε χρήση το άρθρου 5. Τώρα για την προπαγάνδα. Ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρξει χειραγώγηση της κοινή γνώμης. Το δείχνει και η ευρωπαϊκή ιστορία. Δείχνει. Είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένας κόσμος που να πείθει όσους κατοικούν σε αυτόν ότι πρόκειται για την πραγματικότητα ενώ δεν πρόκειται. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική η στρατηγική επικοινωνία. Όχι απαραίτητο για να γίνει μια αντιπροπαγάνδα. Όχι, όχι. Αν μπορεί κανείς να βάλει την αμφιβολία στα μυαλά του κόσμου ότι η προπαγάνδα που ακούνε κάθε μέρα μπορεί να μην είναι αληθινή ακόμα και έτσι θα πετυχαίναμε το στόχο μας. Και για τις κυβέρ. Αν γίνουν θύματα ταυτόχρονα πολλών χωρών κυβερνοεπιθέσεων. Αυτό το θέμα που είναι εδώ, που υπάρχει εδώ είναι η πρόληψη, η αποτροπή και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει μεγάλη σύνδεση μεταξύ μας. Γιατί ξέρουμε ότι πάντοτε ο πιο αδύναμος κρίκος θα καθορίσει τελικά το αποτέλεσμα. Αυτό είναι μήνυμα και για χώρες που είναι πιο προχωρημένες από άλλες. Build walls that are high enough uh, to protect them. Και δεν μπορούν να χτίσουν υψηλά τείχη για να προστατευτούν. Η συνεργασία λοιπόν, οι συμμαχίες ακόμα και με τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι σημαντικές. Σήμερα υπάρχουν 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι online. Σε μερικά χρόνια θα είναι πέντε. Και η διαφορά θα γίνει από τον τώρα αναπτυσσόμενο κόσμο. Εφόσον βέβαια τα δίκτυα είναι ασφαλέστερα. Αυτοπροστασία είναι το θέμα. Επειδή είμαστε πιο συνδεδεμένοι πριν είμαστε και πιο ευάλωτοι. Λοιπόν, αν πολλές χώρες ταυτόχρονα λοιπόν γίνουν θύμα επιθέσεων Υπάρχει η εργαλειοθήκη που μπορεί να οδηγήσει και στην εφαρμογή του άρθρου 5. Μια κυβερνοεπίθεση μπορεί να οδηγήσει στο άρθρο 5. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στην Ένωση χωρίς άρθρο 5. Τώρα για το ρόλο της Ένωσης για την προώθηση στενότερης συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών πληροφοριών. Αυτά είναι θέματα εθνικά, εθνικής κυριαρχίας. Uh, e there is Υπάρχει συνεργασία υπηρεσιών πληροφοριών στην Ένωση, αλλά πάντα μπορεί να βελτιωθεί. Πάντα. Πάντα. Πάντα μπορεί κανείς να πει δεν είναι αρκετό, δεν είναι αρκετό. Αν λοιπόν οι χώρες θεωρήσουν ότι έχουν συμφέρον και όσες έχουν περισσότερες πληροφορίες και οι άλλες έχουν διότι έχουν συμφέρον να συνεργαστούν θα υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία. Αν θεωρήσουν ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών τη χάνουν απαρκούς προστασίας θα υπάρξει επαρκής προστασία. αν τα έθνη καταλάβουν ότι μπορούν να ωφεληθούν από αυτή τη συνεργασία όχι μόνο ως προς τη χορήγηση πληροφοριών αλλά και αναλύσεων και συστάσεων και προσοχής και στήριξης από τις άλλες χώρες τότε θα αυξηθεί η όρεξή τους θα ανοίξει η όρεξή τους για μεγαλύτερη και περισσότερη συνεργασία. Υπάρχουν βέβαια και δυσκολίες. Υπάρχουν δυσκολίες για την ε, χορήγηση εμπιστευτικών πληροφοριών από μια χώρα στην άλλη, αλλά καιρός είναι να αρχίσει μια τέτοια συνεργασία. να υπάρξουν κοινέ πληροφορίες για τον ΝΑΤΟ και την Ένωση. αν κάθε έθνος δεχτεί να χορηγείται τις πληροφορίες θα έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα μπρος. Μπρος. Οι βέλτιστες πρακτικές τώρα και η ανταλλαγή τους δέστε πόσο αποτελεσματικό θα ήταν να συνεργαστούμε ακόμη και με τους εφήβους όπως έγινε για την περίπτωση πολλές φορές επιθέσεων του λεγόμενου Ισλαμικού κυράτους. Πώς να αντιμετωπίσουμε δηλαδή την αγωνία κοινοτήτων που θεωρούν ότι την χάνουν επίθεσης, ε, μυσαλλοδοξία, τέτοια πράγματα πολύ ανάγκη υπάρχει για πολύ στενότερη συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών. Και αυτό είναι κάτι που μας αφορά άμεσα, δεν είναι κάτι μακρινό στη Συρία και το Ιράκ και στους δρόμους της Ευρώπης γίνεται αίμα. Τα παιδιά μας σκοτώνονται και πολλές φορές πηγαίνουν και γίνονται τζιχαδιστές. Άντε, ας σταματήσω εδώ. Ευχαριστούμε, Διευθυντά. Και τώρα κύριο Ρίκ Βάιλς. Thank you, uh, Chair. Um, well, I would maybe not answer all, all the questions because I, I... Πού να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις. Έτσι κι αλλιώς δεν απευθύνθηκαν σε μένα. Αλλά τώρα όσον αφορά τον ορισμό του υβριδικού, ναι, αλήθεια σας λέω, ναι. νομίζω ότι θα ήταν χάσιμο χρόνο οι οργανισμοί αυτοί να προσπαθούσαν να τα βρούνε όσον αφορά έναν γενικό ορισμό. Γιατί άμα τα συμφωνήσουμε ας πούμε, στο ΝΑΤΟ, αυτό δεν να πει ότι μπορεί να τα βρούμε για να έχουμε τον ίδιο ορισμό και στην Ένωση. Ακριβώς αυτό είναι και το πρόβλημα. Άλλο πρόβλημα τώρα, όπως ίσως τα ξέρετε. Οι μετέπειτα ενέργειες των οργανισμών ίσως έχουν να κάνουν με τους ορισμούς και να εκπηγάζουν αυτούς δηλαδή για το πώς θα διατεθούν κάποιοι πόροι για του τι είδου δαπάνες και χρηματοδοτήσεις θα γίνουν αργότερα. Ανάλογα επομένως με το τι κανένας ε, βάζει μέσα στον ορισμό, τι καλύπτει ο ορισμός. Όμως νομίζω ότι το το υβριδικό, αν ανοίξει κανείς ένα λεξικό θα δείτε ότι υβριδικό είναι κάτι το ετερογενές λένε τα λεξικά δηλαδή συνδυασμός διαφορετικών στοιχείων αυτό τι πάνε να πει ότι όπως σας είπα η σύγκριση με ένα μικρόβιο με έναν ιό είναι εύστοχη ότι δηλαδή μεταλλάσσεται συνέχεια δεν έχει την ίδια μορφή συνέχεια το υβριδικό όπως και ο ιός της γρήπης Πάντως, με προβληματίζει το παραδοσιακό πρόβλημα. Τι γίνεται με τον προηγούμενο πόλεμο, πώς αυτό θα το χειριστούμε. Και αυτό μας βοηθούσε στη χώρα μου, δηλαδή ότι πώς θα γίνει να προετοιμαστούμε για έναν πόλεμο που ποτέ δεν έγινε. Υβριδική απειλή. Τι είναι είναι κάτι που εξαρτάται από το πότε κανείς διαβαίνει το κατόφλι της εχθρικότητας, της εχθρικής ενέργειας και οπότε θα πρέπει αυτό να γίνει, να διαβεί κανείς το, το, το με κάποιο τρόπο αισθητό. Α, αυτό όμως δεν ισχύει σε κάθε περίπτωση. Ναι, θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες οι πληροφοριών Πάντως, κάποια κράτη έχουν μεγαλύτερε τεχνικές δυνατότητε από άλλα και επίσης μπορούν να διαπιστώσουν καλύτερα τι γίνεται. Τι γίνεται επί, τόπου. Να έχουν εικόνα, ε, να είναι στρατηγικού επίπεδου οι πληροφορίες που αντλούν. Και είναι και θέμα ασφάλειας πληροφοριών και αντίληψης του πώς η μία υπηρεσία πληροφοριών βλέπει την άλλη. Γιατί αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, πώς να μοιραστούν τις πληροφορίες. Οπότε έτσι υπονομεύονται οι προσπαθίες μας. Τώρα σαν αφορά τις στρατηγικές επικοινωνίες, εμείς συμβάλλουμε στο κέντρο αριστείας για στρατηγικές επικοινωνίες. Οπότε και εδώ είναι το ζήτημα του πώς θα επισημανθεί ένα πρόβλημα, πολύ σημαντικό και αυτό. Όπως είπε δεν είναι όλα παράνομα στην δημοκρατική κοινωνία. Οπότε δεν είναι παράνομο. Και το να στέλνει κανείς επίτηδες λάθος πληροφορίε. στο θέμα σε τι κλίμακα θα γίνεται αυτό, η ένταση του μηνύματος που στέλνει κανείς και κατά πόσον αυτό κρύβει μήνυμα επιθετικότητας, εχθρότητας. Ας το δούμε έτσι σαν ένα τρίγωνο. Οπότε μπορείτε να διαπιστώσετε πού έγκυται το πρόβλημα πλευράς προπαγάνδας. Ένταση, κλίμακα για την ε, εχθρική ενέργεια, όλα αυτά το λένε μπούσουλα για το τι θα κάνει κανείς περαιτέρω. Οπότε ούτε κρατικός ούτε μη κρατικός ε, φορέας, ούτε κράτος ούτε, ούτε άλλο νομικό πρόσωπο του δικαίου θα χρησιμοποιήσει τους πόρους που έχει, τα μέσα που έχει, χωρίς λόγο για να δημιουργήσει ε, κάτι αρνητικό, κάποιο πρόβλημα ε, σε άλλο κράτος ή σε άλλο φορέα. Πάντα κάτι κρύπτει πίσω από τέτοιες ενέργειες. Σας ευχαριστούμε λέει πρώτος τώρα. Θα δώσω το λόγο μόνο σε έναν βουλευτή γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ο κύριος έλεγε λοιπόν να πει το λόγο και θα ήταν ε, καλό να απευθυνθείτε σε ένα συγκεκριμένο άτομο, σε ένα συγκεκριμένο πανελίστα για το ερώτημά σας. Γιατί δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Έχετε το λόγο. Ε, πολύ ευγενικό εκ μέρους Και πολύ λυπάμαι γιατί και οι τρει ενδεχομένω να έχουν να απαντήσουν, αλλά θα, απαντήσουν, θα αποφασίσουν οι ίδιοι. Αν συγκρίνουμε τώρα τι υβριδικές συγκρούσει του παρελθόντος Επιθέσει σε, κυβερν... σε υβριδική βάση. Η Γεωργία ήταν μάλλον ε, αυλαβής, αλλά και πάλι ήταν επίθεση του κράτου. Εδώ πέρα μετά πάμε στην Ουκρανία, όπου... Oh. Η Ισραηλινοί στην τελευταία στην έδρια του Τελαβίβ ε, ρώτησαν τους Ρώσους τι γίνεται για θέματα με διάδοση. Και ύστερα, σε ό,τι αφορά την επίθεση της Βορείου Κορέα στην ε, οικονομική αγορά, στη χρηματοπιστική αγορά της Νοτιού Κορέα, The Middle East. My, my, my question was not... Και κοιτώντας τι έγινε και στην Μέση Ανατολή. Καταλαβαίνουμε φυσικά το θέμα της απειλής, αλλά πέρα από την κατανόηση της απειλής, πώς θα κατηγοροποιούμε αν έχουμε ένα άρθρο 1 και θέλουμε να ορίσουμε το επίπεδο αντίδρασης. Υπάρχει οποιαδήποτε απόπειρα να κατηγοριοποιηθεί το επίπεδο κλιμάκωσης γιατί οι επιθέσεις εγκληματιών στην, από και από τη Λευκορωσία εναρχιστρωμένες κατά πάσα από τη Ρωσία στην ε, Ουκρανία υπάρχουν άμεσες ε, σχετικά ενδείξεις ε, εμπλοκής και των κρατικών αρχών μπορεί και όχι ρωσικών και στην Ουκρανία υπήρξε ανάμειξη των παραδοσιακών στρατιωτικών μέσων και των υβριδικών μέτρων. Και ύστερα στην Κορέα είχαμε απόλυτη επίθεση, στεγνή επίθεση στην χρηματοπιστωτική αγορά. Πιο πολύ από τον τομέα της κατασκοπίας και των δημοσίων υπηρεσιών. Είναι σημαντικό λοιπόν το θέμα του άρθρου 5, το θέμα του πώς κατηγοριοποιούνται αυτές οι επιθέσεις για να αποφασιστούμε, να αποφασιστεί μετά και η αντίδραση. Υπάρχει οποιοδήποτε απόπειρα στο ΝΑΤΟ, στα κρατημέλη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μια τέτοια κατηγοριοποίηση. Or, um, the level of reaction would it be... Ε, και αυτό ασφαλώς θα καθορίσει και το επίπεδο της αντίδρασης. Αυτό πιστεύω θα ήταν ενδιαφέρον για μας. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρος, νομίζω ότι θα πρέπει να αποφασίσουν, και οι τρεις πανελίστε ποιος θα απαντήσει. Και οι τρεις μπορούν να. Εγώ θα απαντήσω επιγραμματικά με μία πρόταση. Το βήμα που κάναμε στο ΝΑΤΟ είναι ότι αναγνωρίσαμε ότι η βρετική αυτή επίθεση μπορεί να αποτελέσει επίθεση βάση άρθρου 5. Δεν έχουμε ορίσει, ούτε έχουμε επιχειρήσει να ορίσουμε το επίπεδο, το όριο. Τι είδους και τι επίπεδου επίθεση μπορεί να αποτελέσει επίθεση βάση άρθρου 5. Αλλά για να σας δείξω πόσο ενωμένοι είμαστε στις προσπάθειές μας, θα τα αφήσω στον συνάδελφο από την Ευρωπαϊκή Ένωση να απαντήσει που δούλευε παλιά και στον ΝΑΤΟ και ήταν εκεί υπεύθυνος για θέματα. Ναι, συντομία για το όριο, για το επίπεδο. Δεν έχει γίνει οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια και ούτε θα γίνει, πιστεύω, στο μέλλον. Και ακόμα και την τρομοκρατία, μετά την 11η Σεπτεμβρίου, όταν έχασαν τη ζωή τους 3.000 άτομα, ξέρουμε ότι χρησιμοποιήθηκε το άρθρο 5 στη συνέχεια. Σημαίνει αυτό ότι στο μέλλον οποιαδήποτε τρομοκρατική επίθεση που θα έχει ως συνέπεια να χαθούν 3.000 ε, ζωές θα έχει ως συνέπεια την κινητοποίηση του άρθρου 5. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Αυτό το θέμα της, ε, του ορίου. Αυτό στέλνει το μήνυμα τι. Ότι αν ε, χαθούν 3.000 ζωές από αυτό το σημείο και πέρα, χρησιμοποιείται το άρθρο 5. Δηλαδή, άμα χαθούν 2.500 ζωές, δεν θα συμβεί τίποτα. Είναι δύσκολο λοιπόν να βάλουμε τέτοια όρια. Το βασικό μήνυμα είναι ότι δεν το κάνουμε, μην το κάνετε γιατί ενδεχομένω να βρεθείτε αντιμέτωποι με το άρθρο 5 ή με μια οποιαδήποτε άλλη πολύ σκληρή αντίδραση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, όχι, δεν υπάρχει καμία τέτοια προσπάθεια. Επειδή είναι και πολύ διαφορετικός ο χαρακτήρας των επιθέσεων ανάλογα με τις ε, ε, συνθήκες. Αυτό εξαρτάται και από το κράτος μέλος, ε, αν μιλάμε για μέλος του ΝΑΤΟ, ε, για το πόσο αξιολογεί κάθε κράτος μέλος την κατάσταση. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε, οποιοδήποτε αυτοματισμός ότι αν υπάρχει τέτοιου είδους βλάβη θα υπάρξει ή τάδε τύπου αντίδραση. Ούτε νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει, θα υπάρξει στο μέλλον, γιατί θα μας αυτό στην αντίδρασή μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ που θέσατε και το ερώτημα. Πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Θα ήθελα να πω το εξή. Για ένα κράτος ε, έθνος, το άρθρο 5 και το όριό του αντικατοπτρίζεται στο αίσθημα που επικρατεί στο έθνος αυτό. Η εξωτερική πίεση το αίσθημα του κατά πόσον βρισκόμαστε υπό επίθεση. Η πρωτοβουλία αυτή δεν προέρχεται από το ΝΑΤΟ, από τη Συμμαχία, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ερωτιέται οι εξωτερικοί παράγοντες αν είναι υπό επίθεση το κράτος. Το έθνος από μόνο του αισθάνεται ή δεν αισθάνεται απειλούμενο. Οι σύμμαχοι αποφασίζουν από εκείνο το τι θα γίνει. Και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να αναλύεται η πραγματική απειλή, η πραγματική επίθεση. Αν μιλάμε για επίθεση με τάγκς, είναι διαφορετικό φυσικά το θέμα των ευρετικών επιθέσεων ωστόσο. Επειδή ακριβώς είναι ασαφές, επαφείται στις χώρες να έλθουν στο ΝΑΤΟ, να έλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πούν ότι κοιτάξτε, είμαστε υπό επίθεση και αυτές είναι οι ενδείξεις, αυτά είναι τα αποδεκτικά στοιχεία. Είναι λοιπόν σημαντικό να γίνουν όλα αυτά Σωστά. Και εδώ είναι σημαντικό οι αντίπαλοι μας, οι εχθροί μας, να ξέρουν ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε βεβαιότητα σε σχέση με την αντίδρασή μας. Ε, και πιστεύουμε ότι οι δύο οργανώσει θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές η προς την άλλη. Η Πρόεδρος. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων καταδεικνύει τις απόψεις ε, και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών και ότι ουσιαστικά υπάρχει καλός συντονισμό. Έτσι κλείνει πολύ ωραία και πολύ ενθαρρυντικά αυτό το σημείο στην ημερησία διάταξη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εξαιρετικούς μας πανελίστες, καθώς και όλα τα μέλη που συμμετείχαν στη συζήτηση. Και σας ευχαριστώ και περνάμε άμεσα στο επόμενο θέμα. Αλλά θα ήθελα καταρχάς να αποχαιρετήσω τους προσκεκλημένους μας. Ladies and gentlemen, please be seated. Καθίστε κυρίες και κύριοι, λέει η Πρόεδρος, διότι ευθύ αμέσως θα προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Και το θέμα είναι η Ευρωπαϊκή Χωροφυλακή. Στην υπηρεσία της ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Έχουμε εδώ τον συνταγματάρχη Ρίο, Φιλίπ Ρίο, που είναι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Χωροφυλακής. Οπότε θα κάνουμε μεταλλική απόφαση μαζί του για να μας εξηγήσει ακριβώς τι προγραμματίζεται, τι προβλέπεται για την Ευρωπαϊκή Χωροφυλακή. Φαντάζομαι ότι αυτό θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Καλώς ορίσατε. Κύριε Συνταγματάρχα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε και κύριοι βουλευτέ. Θα αρχίσω κατευθείαν με την ουσία. Γιατί οι ερμηνείς υφίστανται έναν μαραθώνιο που θα ήθελα να τον ελαφρύνω. Η ανταλλαγή αυτή απόψε, κυρία Πρόεδρε, έρχεται αμέσως μετά την ανάλυση σας για τον υβριδικό πόλεμο, διότι οι δυνατότητες των αστυνομικών και διοκτικών αρχών μπορεί να είναι, μπορούν να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση αυτών των τέτοιων εξωτερικών κρίσεων έτσι ώστε να αναλαμβάνουν ε, το ταχύτερο δυνατόν τη σταθεροποίηση ζωνών κρίσης έξω από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και να συνδυάσουν τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού χώρου ολόκληρου. Μίλησα για έξω από την Ένωση αλλά και μέσα βέβαια και μέσα ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι και οι απειλές επί των συμπολιτών μας. Περνάω τώρα στα αγγλικά, που είναι η γλώσσα εργασίας της Ευρωπαϊκής ε, Χωροφυλακής. και της οποίας ηγούμε από το καλοκαίρι. Ο στόχος ήταν να γίνει μια δήλωση προθέσεων το 2004. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στον ιστότοπο που έχουμε. Πρόκειται για ένα σύντομο έγγραφο. για τη συγκρότηση της ε, χωροφυλακής, ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις δυνατότητες όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια. Και να έχει χαρακτήρα ευρωπαϊκό αυτό το σώμα. Επίσης, θεωρήσαμε ότι έτσι καλύπτουμε και τον χώρο αλλά και τις πολιτικές ασφάλειες και δικαιοσύνης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να σταθεροποιηθούμε και τη γειτονιάζουσα περιοχή και επίσης να συμβάλλουμε και στην ασφάλεια της Ένωσης. Oh, Βλέπουμε τι πίεση υπάρχει στα σύνορά μας την σημερινή ημέρα. Έχουμε κόσμο που έρχεται από άλλες χώρες. Βέβαια, είμαστε νέο σώμα, υπάρχουν και άλλες ε, και που θα κατατείνουν στο να χαλαρώσει αυτή η πίεση στα σύνορα της Ένωσης εάν αυτές οι δυνάμεις αναπτυχθούν σωστά βασική στόχη τώρα. Να υπάρχει ε, κάποια δυνατότητα εκτέλεσης αποστολών αστυνομικού χαρακτήρα όταν υπάρχει κρίση. Να υπάρχει επομένω επιχειρησιακή δομή σε σχέση με κάποια κράτη που θέλουν να βοηθήσουν και γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι καλοδεχούμενη συνεργασία με άλλες ε, ομόλογες, με εμάς δυνάμεις για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Ε, επίσης, ε, ε, έχει συγκροτηθεί έτσι η χωροφυλακή ούτως ώστε να συμμετάσχει σε κάποιες άλλες πρωτοβουλίες ε, διεθνών οργανισμών ΝΑΤΟ, Ηνωμένα Έθνη και άλλου είδους οργανισμούς ή σε κάποιο είδους ad hoc συνασπισμό και έχουμε μένω σε αυτή την ε, δήλωση προθέσεων, ούτως ώστε να προχωρήσουμε σε κάποιο είδους ε, επιχειρησιακό εργαλείο, το οποίο να είναι εκ των προτέρων οργανωμένο για να πετύχει αυτούς τους στόχους. Οπότε αυτό που θέλαμε είναι να υπάρχει ένας τέτοιος οργανισμός, όπως είπαμε προοργανισμένο, εύρωστος και να είναι εδώ να αναπτυχθεί ταχαίως. Το δε αποτέλεσμα είναι ότι μπορούμε να είμαστε και κάτι σαν μία δύναμη ε, γέφυρα μεταξύ κάποιες ε, στρατιωτικού χαρακτήρα επιχείρησης της διεθνούς κοινότητα. σε σχέση με την ε, πολιτικού χαρακτήρα αποστολή που θα μπορούσε να ε, εκτελέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση οπότε έτσι καλύπτεται αυτού του είδους το κενό το οποίο έχει πάρα πολύ ευαίσθητο χαρακτήρα. Πάμε παρακάτω. Τώρα, συγκροτείται ε, το σώμα μας από 7 κρατημέλη. Όλα αυτά έχουν κάποια εθνική χωροφυλακή. Επόμενη διαφάνεια. Βλέπετε τώρα ποια είναι αυτά τα μέλη. Ε, χωροφυλακή, δηλαδή αστυνομικό σώμα με παραδοσιακή αρμοδιότητα αστυνομικού χαρακτήρα και 95% της δραστηριότητας αυτές οι δυνάμεις ε, είναι χαρακτήρα εσωτερικού στη χώρα τους και ας Και έχουμε 360.000 αστυνομικούς για την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας. Οπότε έχουν τις ε, ε, δεξιότητες για την αντιμετώπιση των κρίσεων. Οπότε όλοι αυτοί είναι σε ετοιμότητα για την ασφαλεία μας. Επίσης, υπάρχει και στατιωτικό καθεστώς και παράδοση, ότι δηλαδή αυτοί οι αστυνομικοί ε, μπορούν να αναπτυχθούν για, σε περιπτώσεις κρίσεως και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και σε στατιωτικές επιχειρήσεις. Επίσης, πέραν αυτών των κρατών μελών, έχουμε ε, ένα κρατος μέλος που είναι ε, παρατηρητής. Έχει αστυνομία με στρατιωτικές αρμοδιότητες και εκτελεί 95% της δραστηριότητας στο εσωτερικό. Δεν έχουν επομένω αστυνομική πείρα, οπότε δεν μπορούν εύκολα το know-how που έχουν τεχνογνωσία που έχουν να την αναπτύξουν σε τρίτες χώρες. Και για τον παρατηρητή ισχύει το ότι είναι χώρα υποψήφια που έχει χωροφυλακή. Είναι η Τουρκία. Η Τουρκία είναι παρατηρητής. next slide, thank you. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ταχαίως για να έχουμε χρόνο για ρωταπαντήσεις και συζήτηση. Ε, Εδώ μπορείτε να δείτε τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Χωροφυλακής. Η προστιθέμενη αξία, η μία από αυτές, είναι ότι συνδυάζει τις δυνατότητες της παραδοσιακής της αστυνομίας και τη δυνατότητα να μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα περιβάλλον εχθρικό. Οπότε έτσι μπορεί να έχουμε ένα φάσμα πολλών διαφορετικών λειτουργιών αστυνομικού χαρακτήρα. Τα βλέπετε. Δεν ξέρω αν μπορεί να διαβάσετε αυτά τα γράμματα, τουλάχιστον τα έχετε. Έχετε το, την παράσταση. Οπότε μπορεί έτσι το σώμα μας να πανέβει σε κάποια πρώιμη φάση κρίσης, να βοηθήσει στην προστασία πολιτών και να έχει αστυνομικές αποστολές. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Όταν η κατάσταση βελτιώνεται, βοηθούμε πάλι σε πρώιμη φάση για τη δημιουργία δυνατοτήτων των ε, δυνάμεων ασφαλείας. Και είναι στην κατάλληλη θέση ο κατάλληλος άνθρωπος. Ποιος άλλο το κάνει αυτό καλύτερα. Πώς δηλαδή κανείς μπορεί να έχει αστυνόμευση στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Άρα μπορούμε να ασκήσουμε ε, λειτουργία ιδιοκτικής αρχής, αλλά όσο πιο νωρίς μπορούμε να δημιουργήσουμε δυνατότητες αστυνομικές, τόσο το καλύτερο. Όσο νωρίτερα τόσο μπορεί και να ολοκληρωθεί η αποστολή και να έχουμε εξοικονόμηση χρόνου, ε, χρημάτων κλπ. Αργότερα, όταν η κατάσταση είναι πιο ε, ήσυχη, τότε μπορεί κάποιος από τους εταίρους μας να βοηθήσει για μεταρρυθμίσεις στη, στις υπηρεσίες ασφαλείας. Έχουμε 300.000 εμπειρογνώμενες, οπότε στα πλαίσια της κοινή ε, πολιτικής ε, της ασφάλειας μπορούμε να βρούμε αυτόν που χρειάζεται. Λέτε πρέπει να βρεθεί ο άνθρωπος που να μιλάει τη σωστή γλώσσα. πούμε θέλουμε κάποιον για το Μαλί, αλλά πρέπει να βρούμε κάποιον από γαλλόφωνο περιβάλλον για να πάει στο Μαλί κλπ. κλπ. Τώρα, όσον αφορά το να μπορούμε να καλύψουμε ένα ευρύ φάσμα διαφόρων καταστάσεων, η χωροφυλακή μπορεί να θεωρηθεί ότι ακριβώς μπορεί να λειτουργήσει σαν γέφυρα που σας είπα προηγουμένως. Επόμενη διαφανή. Εδώ βλέπετε είναι παραφορτωμένη αυτή η παράσταση, αλλά μπορεί να δείτε τι έχει γίνει από τότε που συγκροτηθήκαμε. Ξεκινήσαμε με την επιχείρηση U4 Αλθέα. Εδώ υλοποιήθηκε η αρχή της ε, ολοκληρωμένης αστυνομικής μονάδας. Πρόκειτο για κάποιες ομάδες, δημιουργίες ή για μεμονωμένους ε, ειδικού και προγνώμους. Όλοι αυτοί επομένω συναπετέλεσαν μία μονάδα για θέματα δημόσιας ασφάλειας. και έτσι υπήρχε η εμπειρογνωμοσύνη που χρειάζεται. μπορεί να, αυτό μπορεί να αφορά συλλογή πληροφοριών, κατάρτιση, ε, επιχειρήσεις Οπότε είδαμε πως αυτή η αρχή της ολοκληρωμένης μονάδας υλοποιήθηκε. Επίσης, ε, είχαμε και άλλες τέτοιες επιχείρησεις παρακάτω. Ε, είχαμε ταχύτατη ανάπτυξη εκεί στις γαλλικές αντίλες. Υπήρχε μια μονάδα ε, γαλλική, μια ιταλική και κάποιοι κομμάντος Ισπανοί που αναπτύχθηκαν εκεί ταχύως. Στο Αφγανιστάν τώρα, στα πλαίσια του ISAF, εκεί ε, αναπτύξαμε πάνω από 400 ε, αστυνομικούς, τόσο ώστε να φτιάξουμε ε, ένα περιβάλλον ασφαλέστερο από ό,τι υπήρχε. Να βοηθήσουμε την τοπική αστυνομία επιτόπου, στα παζάρια, στους δρόμους. Αλλά αυτό για να το κάνουμε θα έπρεπε να μπορέσουμε να έχουμε και συνεργασία με το πεζικό. Γιατί σε τέτοιο περιβάλλον ήμασταν κάπως έξω από τα νερά μας. Άρα ήμασταν σε στάση, σε θέση αυτοάμυνας. Άρα θα έπρεπε να έχουμε τη βοήθεια για να μην είμαστε έτσι στριμωγμένοι και να υπάρξει το περιθώριο για μια τέτοια επιχείρηση. Αυτά λοιπόν ήταν ε, τρομερές εμπειρίες, πολύ σημαντικές. Παρακαλώ. Αναπτυχθήκαμε στα πλαίσια του U4 RCA πέρσι. Και εκεί εκμεταλλευτήκαμε αυτό που μάθαμε στο Αφγανιστάν. Άρα, αυτό που θέλαμε είναι να δημιουργήσουμε ασφαλείς συνθήκες για τον πληθυσμό. Να μπορούν οι μουσουλμάνοι να ξαναγυρίσουν, να ξανανοίξουν τα μαγαζιά τους. Από τις 7 μέχρι τις 2 τα ξημερώματα ε, δουλεύαμε. Και επίσης ξέραμε ότι σε δύο χιλιόμετρα υπήρχε δυνάμεις πεζικού που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Και όχι ήμασταν υπό την απειλή αυτομάτων. Μετά είχαμε κάποιες ε, πολιτικού χαρακτήρα επιχείρησης. το Μαλί για συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση και, και θα συνεχιστεί και φέτος το καλοκαίρι. Μετά ε, είχαμε επιχείρηση στο Αφγανιστάν, οπότε ακόμα έχουμε αναπτύξει και έχουμε αναπτύξει και βρίσκονται εκεί ακόμα 70 ε, αστυνομικοί. Επίσης, ένας αστυνομικός είναι στην επιχείρηση Human RCA είναι σύμβουλος του επικεφαλής της υπηρεσίας για δικαιοσύνη, αστυνομία, ασφάλεια και βοηθάει μόνος την τοπική χωροφυλακή τον στείλαμε σε αυτή την Αμερικανική ε, αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού ε, η πόλη, το υπόλοιπο προσωπικό είχε φύγει γιατί θέλαμε να δείξουμε ότι στο Μαλί θα συνεχίσουμε τη δράση μας και παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην περιοχή. Τώρα σε παρένθεση σχεδιάζουμε επί πολλούς μήνες το πώς θα γεφυρώσουμε την ε, δράση μας την πολιτική και την αστυνομική. Όμως, ε, επειδή υπήρχε πρόβλημα επιμελητίας, αποσυρθήκαμε από το Μαλί. Τι λέτε, παιδιά. Οπότε μας είχαν υποσχεθεί ε, ενίσχυση επίπεδο επιμελητίας, αυτό δεν γινόταν, θα ήταν πάρα πολύ περίπλοκο μόνοι μας να έχουμε όλη αυτή την ε, αλυσίδα υποστήριξης επιμελητίας, γιατί υπήρχαν και προβλήματα, ε, και προβλήματα επικοινωνίας. Άλλη τώρα δραστηριότητα και αποστολή είναι ο σύνδεσμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ε, υπηρεσία προγραμματισμού στην ε, Λιβύη και εκεί ένας αξιωματικός στην ε, Τίνιδα ούτως ώστε να βοηθήσουμε τον προγραμματισμό και να υπάρχει κάποιος που να συμβουλεύει για την εσωτερική ασφάλεια και βοηθά την υπηρεσία του, των Ηνωμένων της UNSMIL, και, και τις τοπικές αρχές. Επίσης έτσι βοηθούμε τις υπόλοιπες δραστηριότητε για την ε, πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Αυτά για να σας δώσω μια συνοδική εικόνα του τι έχουμε κάνει σε αυτές τις αποστολές και τώρα να τονίσουμε δύο σημεία. Πρώτα πρώτα για την U4RCA και δεύτερον για την UCAP, την ε, επιχείρηση στο Μαλία. Δύο λόγια για αυτές τις ε, μονάδες. Αυτή η μονάδα είχε αποστολή να βοηθήσει το πώς θα σαν ξαναυπάρξει κράτος δικαίου και θα καταπολεμήσει την ατιμορρησία. Γιατί όταν υπάρχει ατιμορρησία έχει πρόβλημα. Ο πληθυσμός και έτσι δεν μπορεί να προστατεύσει κανείς τον κόσμο. Άρα θα πρέπει κανείς να κάνει ό,τι μπορεί κατά των κακών. Uh, two, uh... τη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπιστούν οι εγκληματίες. Οπότε απελευθερώνονται. ή τέλο πάντων ε, τους μεταχειρίζονται δυσανάλογα αυστηρά. Οπότε εμείς προσπαθήσαμε να βρούμε τη μέση οδό. Για αυτές τις ε, μονάδες είχαμε και μηχανικά μέσα και προσπαθήσαμε να ε, βοηθήσουμε όσον αφορά την αποκατάσταση της τάξης και επίσης βοηθήσαμε να ξαναγυρίσουν οι ιδιωτικές δυνάμεις οι στο έργο τους και τις συνεργαστήκαμε μαζί περιπολούσαμε και αυτή η μονάδα είχε και κάποιους ειδικού ε, στην ποινική διαδικασία και βοηθήσαμε και τις τοπικές αρχές σε αυτό το μέτωπο Υπήρχαν και κάποιοι ειδικοί στι υπηρεσίε πληροφοριών που και αυτοί επίσης βοηθήσαν τους τοπικούς ούτως ώστε οι διεθνείς ε, δυνάμεις ασφαλείας να κάνουν τη δουλειά τους και να ενώσουν τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς με το έργο της u Συνέχεια βρήκε συνεργασία με μονάδα του πεζικού, ούτω ώστε να υπάρξει υποστήριξη. Αυτό είναι απαραίτητο όταν κανείς ε, δρά σε τόσο επικίνδυνο περιβάλλον. Και τον πρώτο λόγο τον είχε ή η μονάδα του πεζικού ή οι χωροφύλακες ανάλογα με την κατάσταση. Αν ας πούμε υπήρχε περιπολία σε επικίνδυνη περιοχή. Είχαμε κάποιον από την πολιτοφυλακή της Ισπανίας, είχε πληροφορία ότι κάπου υπήρχε ένα πτώμα στην περιοχή. Οπότε, η μονάδα του πεζικού εξασφάλισε μια ασφαλή περίμετρο και η μονάδα της χωροφυλακής σε συνεργασία με την τόπια αστυνομία πήγαν να ερευνήσουν την κατάσταση για αυτό το πτώμα. Τώρα, κάποια πολύ σημαντικά συμπεράσματα που αντλήσαμε από την επιχείρηση της UFOR. Παρά το ότι χρειάζεται χρόνος για να υπάρχει, να συγκροτηθεί ένα τέτοιο σώμα πολυεθνικό, Ξέρετε, όταν στο Υγείο του έγινε η, σχετική συνδρία, είπαμε ναι, εμεί θα διαθέσουμε αυτή τη μονάδα, οπότε έτσι, έτσι μπόρεσαμε να συγκροτήσουμε αυτό το σώμα, αυτή τη μονάδα. Επίσης, διευκολύνθηκαν οι επαφέ με τον τοπικό πληθυσμό και βοηθήσαμε πάρα πολύ να ε, δράσουν ξανά οι στο δρόμο οι διοικητικές τοπικές αρχές και προστατεύσαμε τους ε, πολίτες. Και ήταν μια πετυχημένη αποστολή. Παρ' όλα αυτά θα ε. μπορούσαμε να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, ιδίως όσον αφορά τη συνεργασία με τους τοπικούς αστυνομικούς, εάν είχαμε ε, προγραμματισμό ακόμα πιο πρώιμο όσον αφορά το τι αρμοδιότητες είχαμε στη φάση του προγραμματισμού της επιχείρησης. Θα πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός ακριβή. προγραμματισμός Συγκεκριμένο. Και αυτό το μάθαμε και τα είπαμε χτε και με τον Γενικό Διευθυντή της ΕΜΕΣ. Άρα είπαμε ότι θα πρέπει στο μέλλον έτσι να προβλέψουμε τον προγραμματισμό μας. Τέλος. Θα ήταν χρήσιμο να υπήρχε συγχώνευση της χωροφυλακής στην Μινούσκα. Ούτω ώστε να υπάρχουν κάποιοι να διεύθυνουν τις πληροφορίες και αυτές τις πληροφορίες να τις αξιοποιούν οι, ε, τα στελέχη μας που δρούσαν εκεί επί τόπου. Αυτή ήταν η Αφρικανική αποστολή Και ξέρετε, το ευρωπαϊκό αυτό στοιχείο εμπλούτησε την αποστολή. Και όταν τελικά κάποιος αποσύρεται, όταν η u εφυγε θα έπρεπε να υπάρξει κάποια στρατηγική εξόδου. Όμως είπαμε ότι σταματάει η στρατηγική λειτουργία, αλλά η λειτουργία της χωροφυλακής κατά τα λοιπά θα είναι ενσωματωμένη στην αποστολή των Ηνωμένων Εθνών. Συνέχισαν να αναπτύσσονται εκεί τα στελέχη μας και αφού τέλειωσε η αποστολή μας συνέχισαν να δρούν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ αλλά όταν ο ΟΗΕ σταμάτησε να παρέχει υποστήριξη μιλητίας τότε αναγκαστήκαμε τους 40 που είχαμε εκεί αναπτύξει να τους ανακαλέσουμε και τους Ισπανούς κομμάντους. Πώς ξέρετε η κατάσταση δεν είναι τόσο εύκολη και ίσως χάθηκε μια ευκαιρία να αναβαθμίσουμε την ε, επιχείρηση του Μινούσκα, της, Μινούσκα τέλος πάντων. So please I know it. Sorry apology. Um, you can see on that chart. λέω γρήγορα και φαντάζομαι ότι στριμώχνω τους ε, διερμηνείς. Βλέπετε τώρα εδώ πέρα σε αυτή τη ε, διαφάνεια τι γίνεται, τι έχουμε κάνει για, για τις επιχειρήσεις στο, στο μπλε κουτάκι, στο μαλλί, και σε επαφή με τις ε, υπηρεσίες του Μαλή. Όλα αυτά αφορούν την εσωτερική ασφάλεια. Βλέπετε σε αυτόν τον πίνακα ότι έχουμε 17 από τους 36 ειδικού ε, τους έχουμε εμείς στη εκεί. Εμείς. Τους ειδικού σε θέματα αστυνομίας ή τους ειδικού αστυνομικούς. Οπότε υπάρχει ε, αυτή η δυνατότητα γιατί έγινε σωστός προγραμματισμός και αυτό έγινε γιατί κινητοποιηθήκαμε και στείλαμε τους καλύτερους μας. Αυτοί πήγαν εκεί στην αποστολή τούτη. Αυτή είναι μια προστιθέμενη αξία. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο όμως. Όλοι γιατί αυτοί είναι οι κανόνες που ισχύουν όσον αφορά την ανάπτυξη των εμπειρογνωμών. Να, δύο παραδείγματα θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο. Να υπάρχει πλήρης τη δυνατότητα τώρα το καλοκαίρι για αυτή την αποστολή και αυτό θα γινόταν αν είχαμε διαφορετικό σύστημα στρατολόγηση. Και του πρώτου μήνε τη επιχείρηση θα μπορούσαμε να έχουμε όλε αυτέ τι θέσει να τι έχουμε ε, γεμίσει με άτομα και μπορούσαμε να αναπτύξουμε αυτούς που χρειαζόντουσαν και τους υπόλοιπους να τους ε, αποσύρουμε. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε το ίδιο καλούς παντού σε κάθε θέση, αλλά εάν υπήρχε ε, κάποιο είδους σωστή μεθοδολογία στη δουλειά μας, θα ψάχναμε τους καλύτερους στην Ευρώπη, οπότε η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να αποδείξει πόσο αποτελεσματική είναι. Και αυτό να γινόταν έγκαιρα. Και να μπορούσαμε να είμαστε σε επιχειρησιακή φάση σε, μέσα σε 6 μήνες. Κατόπιν θα τους αποσύραμε ή κάποιος ανέμενε δεν θα ήταν πια μέλος χωροφυλακής, θα αφορούσε τη συνεργασία με τις ντόπιε αρχές αλλά από την άλλη μεριά η φυσιολογική διαδικασία κρατάει έναν χρόνο. Και εμείς απλώς ε, προσπαθήσαμε να γεμίσουμε τα κενά κάποιο είδους προσωρινή διαδικασία. Έτσι και προχωρήσαμε, αλλά θα είχε σε αντίθετη περίπτωση παραπάνω δυνατότητες η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάθε αποστολή πολιτικού χαρακτήρα. Γιατί στις στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν υπάρχει πρόβλημα, για τις πολιτικές λέμε. Επόμενη διαφάνεια. Δύο λεφτάκια μόνο για την οργάνωσή μας. Interdepartemental. I have a problem of translation between French and uh, I would say. Un comité interministériel. Έχουμε μια διεπουργική επιτροπή υψηλού επίπεδου. Και υπάρχει ε, ο ύπατος εκπρόσωπος του ΙΠΕΞ, ο οποίος συμμετέχει. Επίσης υπάρχει ο διοικητής της χωροφυλακής και επίσης στο οργανόγραμμα υπάρχει και ε, ύπατος υψηλός εκπρόσωπος τέλο πάντων του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης ή της, ε, του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπάρχει μας ένας διπλωμάτης και ένας ε, αστυνομικός και αποφασίζουν τη στρατηγική, την ανάπτυξη. Λοιπόν, αυτή τις αποφάσεις και όταν ρώτησα, μπορώ, θα μπορώ να, να παρατείνω εκεί τη δουλειά ε, στην ομάδα της Λιβύης, Αυτή αποφάσισαν και εάν χρειαστεί να αποφασίζουν κάτι κατεπηγόντως, τότε υπάρχει συνεννόηση η ηλεκτρονική και έτσι αποφασίζουμε ανάλογα με τη σημασία σε κάποιες ε, εβδομάδες ή μέρες. Αλλά θέλουμε να αναπτύξουμε κάποιους και γίνει και κάτι το οποίο έχει δημοσιονομικό, δημοσιονομικές επιπτώσεις. Σήμην είναι αυτή λοιπόν η Διευπουργική Επιτροπή. οποιο εχει δημοσιονομικες επιπτωσεις είμαι διευπουργικη επιτροπη εγω επικεφαλης του στρατηγίου μας και μονίμως στο αρχηγείο μας έχουμε 40 χωροφύλακες. 25 από αυτούς είναι ειδικοί υψηλού επίπεδου. Και αυτοί είναι στην διάθεση της, ε, ε, της πολιτικής για άμυνα και ασφάλεια. Αλλά είπαμε ποιο είναι το έργο μας, δεν είναι αυτό. Βλέπετε εδώ τι μονάδες έχουμε, μπορείτε να το δείτε και στο website και το θέμα είναι ότι θα πρέπει να κάνω εγώ τον προγραμματισμό, πώς θα βοηθήσω μια επιχείρηση της Βρυξέλλες ή κάποια αποστολή. Όποτε κάποιος λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει κάποιο είδους ε, ε, αστυνομικό προγραμματισμό. Οπότε τους πρώτους μήνες μπορώ να αναπτύξω προσωπικό από το στρατηγείο μας το επόμενο. Παρακαλώ. Βλέπετε, εδώ είναι η προστιθέμενη αξία για την ε, κοινή ε, πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Βλέπουμε εδώ πέρα πώς βοηθούμε σε αυτή την ε, ΚΕΠΑ προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλο το φάσμα των αστυνομικών δραστηριοτήτων από την ε, στεναρή ε, υποστήριξη μέχρι και την εκπαίδευση, την παρακολούθηση και την παροχή συμβουλών. Μέχρι και υψηλού επίπεδου μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας. Αυτό πιο γρήγορα από τη οι υπόλοιπες διαδικασίε. Είναι λοιπόν χρήσιμο αυτό μόνο αν η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόσει μια γρήγορη διαδικασία αν δεν χρειάζεται αυτή η γρήγορη διαδικασία, ο συνήθι τρόπο λειτουργία με όλα τα κρατημέλη ε, και με όλου του σχετικού πόρου είναι πιο ορθό από πολιτική άποψη. Αλλά για ειδικέ απαιτήσει σε ό,τι αφορά το χρονικό διάγραμμα και για ασταθή περιβάλλοντα, ε, ίσω ε, να μπορέσουμε να προσφέρουμε κάτι. Είμαστε μία ε, οργάνωση που αποτελείται από πολλούς συντελεστές, όπως σας είπα, και Έχουμε λοιπόν ε, διάφορες μονάδες, έχουμε επιτόπου δυνάμεις, μπορούμε να παρέχουμε ό,τι χρειαστεί, ό,τι χρειάζεται στις κανονικές ε, αστυνομικέ διαδικασίες και δραστηριότητες. Δεν είμαστε σουγιάς ελβετικός, βέβαια. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά τις ικανότητες οικονόμησης γεφυρών. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, αν υπάρχει κάποια πολιτική αποστολή, μπορούμε να δώσουμε δυνατότητα γρηγορότερης ανάπτυξη της. Αν υπάρχει κενό μεταξύ της ε, στρατιωτικής και της πολιτικής αποστολής, μπορούμε να καλύψουμε αυτό το χάσμα και να διευκολύνουμε την ανάπτυξη της πολιτικής αποστολής. Αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένα πίεση, κάποια προβλήματα αναπάντεχα, θα ίσως να είναι λίγο πιο δύσκολο να το καλύψουμε, αλλά μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα τις ανάγκες. Το μόνο πρόβλημα σήμερα είναι ότι η χρηματοδότηση των αποστολών πάντα έχει να κάνει με το μόνιμο προσωπικό και στο αρχή ποτέ δεν προβλέπεται χρηματοδότηση για γρήγορη ανάπτυξη δυναμικού για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όσο δεν προβλέπεται λοιπόν αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε όσο δεν υπάρχει συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Η Eurozone 4 επισέμους ε, δηλώνει ότι μπορεί να αναπτύξει θεωρητικά 800 άτομα προσωπικό μέχρι σε 30 μέρες. Αυτό φυσικά είναι πολύ θεωρητικό και όλα εξαρτώνται από την πολιτική βούληση και το πολιτικό πλαίσιο. Αν υπάρχει όμως μία μεγάλη πρόκληση και μεγάλη βούληση από πλευρά των κρατών μελών, μπορούμε να το πράξουμε αυτό. Μπορούμε να κινητοποιήσουμε δηλαδή τις εμπειρογνώμονες ε, σε ε, όμως έχουμε, εξακολουθούμε να έχουμε το πρόβλημα της αδυναμίας σε ό,τι αφορά θέματα επιμελητίας. Τέλος, ε, κατά πόσον έχουμε δυνατότητα ανάπτυξης ενός συνεκτικού σώματος που θα είναι άμεσα λειτουργικό. Όταν μιλάμε για ένα σώμα από 5-6 κρατημέλη, όχι μόνο από ένα κρατός μέλος, θα έχουν τις ίδιες παραδόσεις θα έχουν τις ίδιες παραδόσεις, θα έχουν τις ίδιες διαδικασίες. Όλοι θα εφαρμόζουν την ίδια μεθοδολογία και τον ίδιο προγραμματισμό. Και άρα μπορούμε να φτιάξουμε μια τέτοια ομάδα σε κάποιες εβδομάδες. Ενώ οι άλλοι εμπειρογνώμονες οι οποίοι έρχονται με διαφορετικές προσεγγίσεις, με διαφορετικές παραδόσεις από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πλούτος αυτός. Δεν αντιλέγω, αλλά παίρνει μήνες για να σχηματιστεί μια τέτοια ομάδα. Για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, λοιπόν, μπορούμε να παρέχουμε μια άμεση, άμεσα λειτουργική τέτοια ομάδα. Στην επόμενη διαφάνεια, αν θέλετε να κοιτάξουμε, να πω για ένα λεπτό τι γίνεται. επειδή δύο χρόνια διαπραγματευόμαστε μια συμφωνία πλαίσιο με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Στο τελική ανάλυση πλέον ε, ε, στέθηκε με επιτυχία αυτή η διαπραγμάτευση, έχουμε το έγγραφο και περιλαμβάνουμε, περιλαμβάνεται το νομικό πλαίσιο της ανάπτυξης ΚΕΠΑ και ότι ισχύουν οι συγκεκριμένοι κανόνες χρηματοδότησης. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σύστημα το οποίο θα προτιμάται σε σχέση με το Eurogent 4 και τις άλλες ε, συνεισφορές. Έτσι λοιπόν μπορούμε να υποστηρίξουμε την ΚΕΠΑ στη διαδικασία προγραμματισμού. Επίσης κοιτάμε το πώς ε, μπορούμε να αναπτύξουμε τις δυνάμεις και την ε, γεφύρωση αυτή. Πώς μπορούμε επίσης να βελτιώσουμε και να εφαρμόσουμε το σύστημα για τις ε, διαγωνισμούς. Στην επόμενη διαβάνεια. Προκλήσει και το τι θα πρέπει να γίνει στο μέλλον. Καταρχά θα πρέπει να εφαρμοστεί το διοικητικό, η διοικητική ρύθμιση και καλό θα ήταν να γίνει αυτό, αλλά αυτό προποθέτει ότι θα συμφωνήσουν όλα τα κρατημέλη, όχι μόνο αυτά που συμμετέχουν στο Eurogent Fork. είναι πάρα πολύ καλό αυτό για κατεπίκουσε καταστάσει όπου υπάρχει μεγάλη έλλειψη ασφάλεια. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν θα μπορούσαμε να παρέχουμε την εμπειρογνωμοσύνη πέρα από την επιλογή, την κανονική, το κανονικό σύστημα επιλογή, το οποίο προαπαιτεί μήνες ασφαλώς και δεν μπορεί να είναι γρήγορο. Και για να αρθούν ε, οι αμφιβολίε των μελών που δεν είναι στο γύρο June Fair, που τι καταλαβαίνουμε και είναι λογικέ, θα πρέπει να κατανοήσουν τα κράτη-μέλη ότι δεν. Ε, να κατανοήσουν τι γίνεται τα κράτη-μέλη που δεν έχουν χωροφυλακή. Επίση θα πρέπει να βελτιωθεί η πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων προκειμένου να υπάρξει καλύτερη, ε, καλύτερο συγχρονισμός μεταξύ PSC και SIMIN. Γιατί μπορεί να ληφθεί η απόφαση δεν μπορεί μάλλον να ληφθεί η απόφαση να συμμετάσχουμε σε διαδικασίε ΚΕΠΑ όσο δεν έχει κληθεί η eurogen 4 από το PSC. Εδώ λοιπόν χρειάζεται καλύτερο ε, ε, προγραμματισμό χρονικό από πλευρά των Βρυξελών. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, κάλυψη των αδυναμιών που έχουμε σε ό,τι αφορά την επιμελητία. Προφανώς, εμείς είμαστε, προοριζόμαστε για να έχουμε αστυνόμευση στη χώρα μας. Δεν έχουμε τόσο μεγάλη εμπειρία για, την, για τις αποστολές. Άρα, αν δεν βρούμε κάποιο μηχανισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη, τη γρήγορη ανάπτυξη και για τη Eurogen 4 ε, ή και για οποιαδήποτε άλλη συμμετοχή άλλου κράτους μέλους. Αν δεν έχουμε υποστήριξη λοιπόν για την γρήγορη αυτή αντίδραση, τα πράγματα δυσκολεύουν ασφαλώς. Τέλος. Έτσι όπως έχει κατάσταση λοιπόν τώρα, σε κάθε περίπτωση καλή είναι η διαχείριση κρίσεων, αλλά πολύ καλύτερη είναι η πρόληψη κρίσεων και αυτό κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε στην Ενησία, όπου χρειάζεται ε, φυσικά έντονη υποστήριξη. Ίσως λοιπόν η Eurogent 4 θα μπορούσε να προσφέρει τα φώτα της και την εμπειρία της για την πρόληψη τέτοιων κρίσεων. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη αν μακρηγόρησα, αλλά νομίζω ότι κάλυψα πολλά θέματα. Η ε, Πρόεδρος τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δαγματάρχη. Ένα αίτημα έχω για ερώτημα. Mr. So thank you very much. Ευχαριστώ πολύ συνταγματάρχα μου. Η γερμανική καμπίνα τουλάχιστον σας μετέφρασε πολύ σωστά και πολύ γρήγορα. Εξ του ΕΛΚ και γενικότερα σας ευχαριστούμε για την προσέλευσή σας. Το 2007 αν το θυμάστε κάναμε την πρώτη μας έκθεση για τις ε, αμυντικές δυνατότητες της Ένωσης. Επισκεφθήκαμε την Ιταλία και δυστυχώς το δικό μου κράτος μέλος είχε μεγάλες αντιρρήσεις γιατί Ξέρετε ότι το σύνταγμά μας απαγορεύει το συνδυασμό στρατού και αστυνομίας. Αλλά θα ήθελα να ξανατονίσω τη σημασία που έχουν αυτές οι δυνατότητες συνδυασμού. Γιατί όποτε χρειάζεται να αυξήσει κανείς τις δυνατότητες τους, του, μια απάντηση θα ήταν αυτού του είδους η Ευρωπαϊκή Χωροφυλακή. Γιατί καμιά φορά και σε περιοχές σειράξεων χρειάζονται αστυνομικές δραστηριότητες. And as Και γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω την προσπάθεια. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, στο τέλος μιλήσατε για συμφωνία ή μεγαλύτερη ολοκλήρωση στην, ε, στον Καπαμά. Και θα ήθελα να ρωτήσω τι αναμένετε Ακριβώς. Τι θα θέλατε ως προς την μεγαλύτερο συνδυασμό και την πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Το κοινοβούλιο μας έγραψε σχετικό έκθεση το 7 Από πρακτικής λοιπόν απόψεως, τι φρονείτε σε υποπολιτικό επίπεδο ως εμπειρογνώμων. Ο κύριος Μπούχνερ. Και εγώ πολύ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που Μα αφιερώσατε το χρόνο για να την παρουσίαση αυτή. Μία σύντομη ερώτηση έχω να σα κάνω. Έω τώρα η κατάσταση δεν ήταν καθόλου δεδομένη. Δεν ήμασταν καν κοντά σε μια τέτοια κατάσταση. Επί της αρχής όμως θα ήταν ε, δυνατόν να εντοπιστεί και να βασιστεί στο ιστορικό της Ευρώπης ε, η Eurogen 4 και έχω υπόψη μου συγκεκριμένα το άρθρο 222 τη συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί της αρχής θα ήταν δυνατό κάτι τέτοιο ή πρόεδρο. Ναι, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη στις ερωτήσει μου. Uh, Στι αρχέ λοιπόν του έτου. Mm. είδαμε Είδαμε λοιπόν την απόδοση της Ευρωπαϊκής Χωροφυλακής και των μελών της αποστολής αυτής. Και τη γενική αντίληψη που ήταν ε, φυσικά πάρα πάρα πολύ θετική. Θα ήθελα να ζητήσω να μας πείτε τι γίνεται με το follow-up, γιατί τότε ήδη υπήρχαν αμφιβολίες και φόβοι που είχαν εκφραστεί. Και θα θέλαμε να ξέραμε, δηλαδή, τι θα πρέπει να γίνει μετά την απόσυρση των δυνάμεων. Κάποια σίγουρα κατάρτιση, εκπαίδευση. Uh, rather difficult, once more rather difficult and, and uh, we face... Uh, Σε ό,τι αφορά δηλαδή την κατάσταση στο Μπαγκέ που είναι πάρα πολύ δύσκολη στο Μπαγκέ, όπως και στο Αφγανιστάν μετά την ναι, ανακατάληψη πέντε μεγάλων πόλεων, ξαφνικά αντιμετωπίσαμε τεράστια προβλήματα. και είμαστε αρκετά απεσιόδοξοι. Αλλά για πείτε μας πώς εκτιμάτε εσείς την κατάσταση. Uh, please. Thank you very much. Uh, uh, the first question, what, what is required to better integrate Eurozone 4? Uh, you have different... Τι χρειάζεται για να εφαρμοστεί καλύτερα και για να ενσωματωθεί καλύτερα η Eurozone 4? Το καλύτερο και το πρώτο τμήμα είναι να υπάρχει καλύτερο σχεδιασμό. Μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση με το να υπάρχει ένα στρατιωτικό σχεδιασμό στη γύρω Gen4. Το στρατιωτικό δεν μα χρειάζεται για να κάνουμε τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό. Αυτό που χρειάζονται είναι προγνωμοσύνη στη χωροφυλακή. Για οργανωθεί ε, e Μπορούμε δηλαδή να, στη Βενιστέντα που είναι η βάση μας, να κάνουμε το σχετικό προγραμματισμό. Ε, ο στρατέος λοιπόν ξέρει τι να κάνει. Το θέμα είναι κατά πόσο θα μας καλέσει εγκαίρω για την πολιτική τώρα, την, την πολιτική αποστολή. Δεν υπάρχει τέτοιος τρόπος ανάπτυξης ε, αστυνομικών δυνάμεων και προγραμματισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει διαδικασία προγραμματισμού, τα σχετικά έντυπα, αλλά δεν υπάρχει κάποια τεχνική στον προγραμματισμό. Για να μας εγγυηθεί καλύτερη, την καλύτερη ανάλυση και τον καλύτερο σχεδιασμό της κατάστασης. Τι θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε και αυτό θα προτείνω είναι να παρέχουμε τις ε, εμπειρογνωμοσύνη μας στο σχεδιασμό συμπληρωματικά προς τις δικές τους ικανότητες προγραμματισμού. Δεν πρόκειται να τα κάνουμε αυτά από μόνοι μας. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε αύριο. Είμαστε έτοιμοι. Δεν σημαίνει η συμμετοχή στον προγραμματισμό ότι στόχος μας είναι να, να αναπτυχθούμε και εμείς στην αποστολή. Όχι. Υπάρχει το σκέλος του προγραμματισμού, υπάρχει το σκέλος της ανάπτυξης δυνάμεων αν αναπτύξουμε και δικέ μα δυνάμει, θέλουμε φυσικά να συμμετέχουμε στον προγραμματισμό και στο σχεδιασμό. Αυτό όμω είναι διαφορετικό. Σε δεύτερο επίπεδο. Τα χρήματα. Οι πόροι. Αυτό δεν αφορά ασφαλά μόνο τη Eurogen4. Αφορά όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν να αναπτύξουν ένα σώμα αστυνομικών. Υπάρχουν λοιπόν μέσα στην ε, Υπηρεσία εξωτερική δράση, στο FBI, που διευκολύνουν το σκέλος αυτό. Το πρόβλημα είναι πώς μπορεί σε πρώτη φάση, στις πρώτες φάσεις του προγραμματισμού να προβλεφθούν οι ανάγκες που θα προκύψουν και να υπάρχουν ε, σωστή πρόβλεψη. Άρα εδώ πέρα συνδεόμαστε με το τρίτο επίπεδο που είναι η πολιτική βούληση. Χρειάζεται μεγαλύτερη εμπλοκή στη φάση του προγραμματισμού. Στο Παρίσι ήμουν ε, υπεύθυνο για την χωροφυλακή και για τη συμμετοχή και τον προγραμματισμό. Για να υπάρξει όμως συμμετοχή των υψηλόβαθμων αξιωματούχων για να κατανοήσουν πώς μπορεί να βοηθήσει η χώρα φυλακή σε περιπτώσεις ε, ανάγκης ήταν πάρα πολύ περίπλοκο. Και για να γίνει κατανοητό αυτό, πραγματικά ήταν μαραθώνιος. Σήμερα, εδώ στις Βρυξέλλες, είμαστε... Υπάρχουν εκπρόσωποι της ΚΕΠΑ. Εδώ στις Βρυξέλλες λοιπόν υπάρχουν πιο πολλοί πρόθεμοι. Περιλαμβάνει αυτό το PSC. Μπορεί να περιλαμβάνει ενδεχομένω και το κοινοβούλιο. Αυτά είναι, λοιπόν τα τρία επίπεδα προετοιμασία. Ε, Προπολογισμό και η πολιτική απόφαση. Για το πώς αναπτυχθεί η Eurogen Force στην Ευρώπη. Και εδώ πέρα επανέρχομαι στην ε, δήλωση του προθέσεων. Η Eurogen 4 είχε ως σκοπό να υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες οργανώσεις στην αντιμετώπιση και διαχείριση κρίσεων. στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο τη Νίκαια το 2002, αν δεν κάνω λάθο, διευκρινίστηκε ότι αυτό ήταν εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ιστορικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί. Υφιστάμενοι. Ενδεχομένω να χρειάζονται βελτίωση. Αλλά σίγουρα η Eurogenfor δεν προορίζεται για εσωτερικέ διαδικασίε. Και επίση δεν εφαρμόζονται και οι συγκεκριμένε ειδικέ τεχνικέ ε, διαδικασίες και δεν πιστεύω ότι αρμόζουν αυτές στην Eurogent 4. Δεν μπορούμε να τα μπλέξουμε αυτά τα δύο. Η προβληματική, η στρατηγική υποστήριξη, η στρατηγική προσέγγιση θα πρέπει να είναι τα ίδια όλα αυτά. Αλλά θα πρέπει να ορίζονται οι διαφορετικοί τομείς με σαφήνεια. Και υπάρχουν ε, και νομικά ένομα μέσα τα οποία χορηγούν τη δυνατότητα μιας χώρας να υποστηρίξει μια άλλη. Και νομίζω ότι υπάρχουν σχετικές διατάξεις. Αυτά λοιπόν μπορεί να επεκταθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά να μην τα μπλέκουμε τη Eurogen Force, παρακαλώ. Γιατί δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας, το, η εντολή μας. When we are deployed there, we are able to keep, once again, I said, the... the, the, uh, Σε ό,τι αφορά τη Μινούσκα, σε ό,τι αφορά τη μουσουλμανική, ε, το μουσουλμανικό πληθυσμό, όταν ε, σχεδόν μιλούσαμε για την οκάθαρση, Τελικά ο κόσμος αυτός επανήλθε, καταστάθηκε και τα πράγματα βαλτιώθηκαν. Αν ε, επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση, θα έρθουν και άλλοι άνθρωποι στις ε, πόρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό επηρεάζει ασφαλώς και τον ευρωπαϊκό χώρο. Και θα πρέπει να βρούμε, να δούμε στην, ε, τι γίνεται με τον ΟΗΕ. γιατί στον ΟΗΕ πάντα υπάρχει το θέμα ότι θα πρέπει να αναπτύξουν τις ίδιες τους ικανότητες. Θα πρέπει να υπάρχουν, ε, να γίνει κάποια αναζήτηση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη δυνάμεων της αστυνομία και του χωροφυλακής του Μαμακό και σε άλλες επαρχίες. Πώς θα γίνει αυτό, υπάρχουν κάποια εργαλεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο, το PSC είναι έτοιμα να αναπτύξουν μια πολιτική αποστολή. Γιατί όχι. Αν όχι, μπορούν να γεμίσουν το χάσμα, το χρονικό χάσμα. Σε ό,τι αφορά την ε, ασφάλεια και την ειρήνη. Και η Eurogent 4 ενδεχομένω να μπορέσει να παρέχει υποστήριξη. Αν χρειαζόμαστε λοιπόν κατεπηγόντω ανάπτυξη τέτοιου δυναμικού στην παρούσα φάση η 4 δεν μπορεί να το κάνει αυτό μόνη της. Αλλά έχουμε άτομα υπεύθυνα για τον πραγματισμό, που σημαίνει ότι μπορούν να δώσουν τα καλύτερα εργαλεία στο εκάστοτε έργο. Και μπορούμε λοιπόν να δώσουμε υποστήριξη και αν υπάρξει πολιτική αποστολή, είμαι βέβαιος ότι επίσης θα είναι δυνατόν Μίλησα για τον Παμακό και για τον Μπάγκη. Γιατί είμαι μεταξύ των δύο αποστολών και καμιά φορά τα μπλέκω. It doesn't need, in, it doesn't need an answer and I don't need in uh, translation. Just a hint. Um, out of the experience there is the, the political... Επί τη βάση της ε, εμπειρίας, τι λέτε, υπάρχει πολιτική βούληση για την οργάνωσης για αυτόν τον τρόπο ή θα γίνει πρώτα πρώτα αυτή η αλλαγή στο έργο σας και κατόπιν θα αναγκαστούν οι πολιτικοί να ακολουθήσουν. Ε, υπάρχει αυτό το πρόγραμμα γιατί θα πρέπει να προσέξουμε να μην υπάρχει ε, αποτέλεσμα, για σαν αποτέλεσμα η εξουδετέρωση της δικής σας δράσης και να μπορέσετε να συμμετάσχετε και να υπάρχει κάποιο πολιτική συμφωνία ή κάποιο είδου μνημόνιο κατανόησης. Και έτσι αυτό το χρησιμοποιήσετε σαν μια εναλλακτική προσέγγιση και να υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, το ερευνητικό πρόγραμμα στα, πλαίσια του ορίζοντος 2020. Να υπάρχει χρηματοδότηση, οπότε και από πολιτικής πλευράς τα πράγματα να έχουν διευκολυνθεί για να μπορέσετε να ενταχθείτε σε αυτό το πλαίσιο. Γιατί αυτό στο παρελθόν ήταν πρόβλημα. Οπότε μπα και έτσι, κοιτάξτε, μπα και έτσι ε, με τις σημερινές σας επαφές μπορέσετε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα και να προχωρήσετε όσον αφορά την ένταξη αυτή. Η πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς θα πρέπει να κηρύξω τη λήξη της συνεδρίασης και θα πρέπει επίσης να ευχαριστήσω τον συνταγματάρχη για την πλήρη παρουσίαση που έκανε. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι που έχετε συμμετάσχει αλλά επίσης να ευχαριστήσουμε και τους ε, διερμηνείς. Και το προσωπικό μας κράτησε λίγο παραπάνω η συνεδρίαση, αλλά ελπίζουμε ότι ήταν ενδιαφέρουσα. Πέρα συνεδρίαση. Sorry. Our next meeting is... Uh, Επόμενη συνεδρίαση, 15, 15 Δεκάτου.